Mm. Nous commençons notre, réunion. Je vous invite à Αρχίζουμε. Αρχίζουμε με τη συνεδρίασή μας. Εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να σας ε, μεταφέρω ορισμένες αλλαγές σε σχέση με την αρχική ημερήσια διάταξη. Χτες η γραμματεία σας απέστειλε την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Καταρχήν θα μας απασχολήσει η τραγική κατάσταση στη Λιβύη και γι' αυτό ζήτησα να προσθεθεί ένα σημείο 6 στην ημερήσια διάταξη όπου θα ζητήσουμε από την Κομισιόν να μας αναφέρει ποια μέτρα έχει λάβει για να βοηθήσει τους πρόσφυγες που βρίσκονται στα σύνορα μεταξύ Λιβύης και την Ισίας. Επειδή οι δύο επιτροπές ΑΦΕΤ και ΝΤΕΒΕ ε, έχουν φορτωμένη ημερήσια διάταξη, θα προσθέσουμε μία ε, πρόταση σύστασης, όπως μας ε, είπε η κυρία Στρίφλερ, θα προσθέσουμε το θέμα της 66ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό δεν θα επηρεάσει την ημερήσια διάταξη, διότι ο κύριος Γκέρενς θα μας μιλήσει παράλληλα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την αρρωγή των τρίτων χωρών. Άρα, στο σημείο 13 θα ήθελα να σας πω ότι η έκθεση Γκέρενς έχει αντικατασταθεί από την έκθεση Στρίφλερ. Επίσης, ε, υπάρχει μια άλλη αλλαγή στο 15 θα μιλήσουμε για το feedback ως προς το δημοκρατικό έλεγχο για τα μέτρα εκτέλεσης του DCI. Θα μας απασχολήσει λοιπόν το θέμα του ασύλου και της μετανάστευσης. Υπάρχουν σχόλια ως προς την ημερήσια διάταξη στη νέα έκδοση που σας απεστάλλει χθες από τη Γραμματεία. Εάν όχι, θεωρώ ότι εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Θα έχετε λάβει τα πρακτικά της 25ης, 26 Ιανουαρίου και 7 Φεβρουαρίου. Εάν έχετε σχόλια θα ήθελα να τα κοινοποιήσετε στη γραμματεία πριν από το τέλος της συνεδρίασης. Αλλιώς θεωρούμε ότι τα πρακτικά εγκρίνονται. Δεν έχω άλλες ανακοινώσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάποια ανακοίνωση προς εμάς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα απλώς να σας ενημερώσω για να σας πω ότι ο Επίτροπος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον Ειρηνικό, όπου θα συμμετάσχει στο Pacific Island Forum και έχει πρόθεση να υπογράψει ένα πρόγραμμα καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών στα πλαίσια μιας περιφερειακής στρατηγικής για τον Ειρηνικό που θα ασχοληθεί, θα αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Κάτι άλλο που θα ήθελα να σας κοινοποιήσω, που ίσως σας ενδιαφέρει, είναι ότι το FID και το Υπουργείο, το Βρετανικό, Βρετανικό Υπουργείο Συνεργασίας έχει συντάξει μία έκθεση σε σχέση με το ΕΤΑ. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει ίσως να βελτιωθεί κάπως το κείμενο. Εν πάση περιπτώσει, η εξωτερική αξιολόγηση του FID είναι πολύ θετική. Αυτά ήθελα να σας ανακοινώσω. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Τώρα, ε, ως προς το έκτο σημείο της ημερήσιας διάταξη, σημείο 6, α, θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή σε σχέση με αυτή την εξαιρετική έκθεση από πλευράς συντηρητικών ως προς την έκθεση του FID. Χρειάστηκε να υπερασπιστώ την ε, Κομισιόν δημοσία και στον Βρετανικό τύπο. Και βλέπω ότι εδώ γίνεται λόγος για τα Funds και τα κονδύλια του ΕΤΑ μέσα στα πλαίσια της ολοκλήρωσης και της υλοποίησης του προγράμματος. Θα πρέπει λοιπόν να το δούμε και σε επίπεδο Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και Επιτροπής Προϋπολογισμών και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να υπεραμεινθούμε αυτή της έκθεση. Ο κ. Μπέρμαν. Επειδή υπάρχουν ε, αγαστές σχέσεις ε, μεταξύ Ντεβε ε, και υφυπουργού Μίτσελ, θα ήθελα να αναθεωρηθεί αυτή η απόφαση να μην χρηματοδοτείται πλέον ο ε, οργανισμός, Διεθνής Οργανισμός Εργασίας. Ο κύριος Μίτσελ αποφάσισε ότι δεν θα πρέπει να την χάνει περαιτέρω, να τύχει περαιτέρω χρηματοδότησης ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας και νομίζω ότι είναι πολύ λυπηρή αυτή η απόφαση της Βρετανικής κυβέρνησης είναι ένα πολύ θλιβερό προηγούμενο. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μία ανταλλαγή απόψεων με τον Υφυπουργό και τον Γενικό Γραμματέα. Λοιπόν, σημείο 6. Τι θα γίνει με τους ε, εκπατριστέντες από τη Λιβύη. Ο κύριος Λούκνερ, θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Λούκνερ από την ΕΚΟ, ο οποίος θα μας πει ποια είναι τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσουμε τους εκτοπιστέντες από τη Λιβύη. Κύριε Λούκνερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, κύριε Σιγητά, εντάχει θα σας πω πώς έχει η κατάσταση όπως την γνωρίζουμε σήμερα το πρωί. Οι συνολικοί εκτοπιστέντες ανέρχονται σε 160.000 από όσο γνωρίζουμε που πέρασαν τα σύνορα με την, Ισία Αίγυπτο και ίσως και Αλγερία και Νίγηρα. Η κατάσταση στην Αίγυπτο είναι κάπως ε, καλή ελεγχόμενη, δηλαδή ο Ερυθρός Σταυρός και η Ερυθρά η Μισέλινος έχουν οργανώσει κάπως τους καταβλισμούς των εισερχομένων. Η πιο σταθής κατάσταση αφορά τα σύνορα Λιβύης την Ισίας, όπου έχουμε μετάβαση 6.000 Αιγυπτίων ημερησίως. Βλέπουμε όμως ότι συνολικά 40.000 παραμένουν στη Λιβύη διότι την Ισία έκλεισε τα σύνορα καθότι δεν υπάρχουν ε, δυνατότητες, ε, ε, δυνατότητες αποδοχής. Και εξαφανίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι, ο Καντάφη απέστειλε τρόφιμα, δηλαδή τα έριξε πάνω από τα τείχη, όμως δεν ξέρουμε ποια είναι η τύχη αυτών των ανθρώπων. Προφανώς θα βρίσκονται σε κάποιο καταβλισμό από λιβικής πλευράς. Αυτή είναι η κατάσταση όπως την γνωρίζουμε για τους 40.000 εκτοπιστέντες στα σύνορα. Από την ισιακής πλευράς έχουμε 15.100 άτομα, αλλά ο αριθμός αυξάνεται στους καταβλισμούς της Τινησίας. Ως προς τη Λιβύη, η κατάσταση προς Ανατολάς, δηλαδή προς τη Βενγάζη, είναι κάπως ε, ήσυχη, όμως δυστυχώς οι μισθοφόροι επιτέθηκαν περίπου 100-200 χιλιόμετρα κάτω από τη Βενγάζη. Η Επίτροπος Γεωργίεβα μετέβη χτες στην Τινησία και κάλεσε, και κάλεσε την κυρία Γιώρη που είναι η Φουπουργός εξωτερικών υποθέσεων να τη συνοδεύσει. Θα παρευρεθούν στα σύνορα για να δουν τι πρέπει να γίνει, σύνορα μεταξύ Λιβύης και Νησίας. Εστιάζουμε την προσοχή μας καταρχήν στη εκένωση των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από όσο γνωρίζουμε 30 Ευρωπαίοι πολίτες έχουν απομείνει που θέλουν να εγκαταλείψουν την χώρα, υπάρχουν και άλλοι χίλιοι που παραμένουν και έχουμε καναδικές πτήσεις προς την Τρίπολη για να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κατάσταση. Στις 22 Φεβρουαρίου στάλει μία ομάδα εμπειρογνωμόνων, τώρα έχουμε δύο εμπειρογνώμονες στην Αίγυπτο, δύο απεστάλησαν χτες στη Λιβύη και τέσσερις στην Τινησία. Επίσης έχει αποσταλεί ένας εμπειρογνώμων με την UNCTAD που μετέβη στην Τινησία χτες. Ως προς τα δελτία τύπου που προκαλούν μεγάλη σύγχυση θα ήθελα να πω ότι οι εμπειρογνώμονες δεν είναι οπλισμένοι και δεν συνοδεύονται. Εμείς θεωρήσαμε ότι δεν θα πρέπει να συνοδεύονται από μία οπλισμένη δύναμη και τώρα συνοδεύονται από τον Ερυθρό Σταυρό. Όπως ανακοίνωσε και ο πρόεδρος Μπαρόζο, αυξήθηκε η αρρωγή σε 10 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, στην ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες δώσαμε 5,5 εκατομμύρια ευρώ και στον Διεθνή Οργανισμό ε, Μετανάστευσης και το ΜΙΓ θα προβεί στην επιμελητιακή βοήθεια προς την ύποτη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες και το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Έχουμε αποστείλει έξι Ευρωπαίους με το ΜΙΚ έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιβλέψουμε την κατάσταση in situ με τις τινησιακές αρχές. Ως προς την δύναμη που έχει μεταβεί προς τα εκεί, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αρχίσει την αποστολή αεροπλάνων και πλοίων για τον επαναπατρισμό Αιγυπτίων που βρίσκονται στην Τινησία αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η δυνατότητα εκένωσης 12.000 ατόμων. Κατά τις επόμενες ε, πέντε ημέρες ο Υπουργός Φρατίνη επίσης τόνισε ότι η Ιταλία θα συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια έτσι ώστε να υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες εκένωσης. Επίσης και άλλα κράτη-μέλη έχουν δώσει έχουν χορηγήσει ανθρωπιστική βοήθεια και από ό,τι γνωρίζω 8 εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί από την Δανία, 660.000 από τη Γερμανία και η Φιλανδία 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Γνωρίζω ότι και άλλα κράτη-μέλη βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία χορήγησης και κινητοποίησης χορήγησης ανθρωπιστικών πόρων. Κύριε Γκέρενς, έχετε το λόγο. Υπάρχουν πολλά... πολλά θέματα, νομίζω, μπορούν να μας απασχολήσουν στην υπόθεση αυτή. Θα ξεκινήσουμε με τα εξή ερωτήματα. Πρώτον, έχετε κάποιον ακόμη με τον οποίο να μπορείτε να επικοινωνείτε σε επίσημο επίπεδο στη Λιβύη. Είπατε ότι συνομιλείτε με ανθρωπιστικές οργανώσεις, με την Ερυθρά Εμισέλινο που είναι το αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού στη Λιβύη, με άλλες ανθρωπιστικές φαντάζομαι οργανώσεις, αλλά μέχρι πού μπορείτε να προχωρήσετε έτσι ώστε να εξασφαλίσετε και διάλογο με τις ε, αρχές της Λιβύης. Γιατί έχουμε δει ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις τέτοιου είδους συνομιλία, επαφή παρέμεινε δυνατή. Εδώ για τη Λιβύη έχω πολλές αμφιβολίες. Και κάτι ακόμη, η χρηματοδότηση και ξέρουμε ότι αυτό στη διάρκεια του έτους θα μας προξενήσει πολλές δυσκολίες. Μήπως λοιπόν αυτή η χρηματοδότηση οδηγήσει τελικά σε μία μορφή αγώνα δρόμου μεταξύ των ποσών που θα χορηγούνται ε, για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης σε χώρες που δεν είναι αναπτυσσόμενες χώρες αλλά αναδυόμενες και ποσών τα οποία θα έχουμε ανάγκη προκειμένου να στηρίξουμε πράγματι τις αναπτυσσόμενες χώρες. Κύριε Μίτσελ. Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Ευχαριστώ την Επιτροπή για τα όσα μας εξέθεσε και χαίρομαι που επισκέπτεται την περιοχή ο Επίτροπος. Είναι μια περιοχή αυτή η οποία πράγματι μπορεί να οδηγήσει σε εξάρσεις, μπορεί τα πράγματα να ξεφύγουν από τον έλεγχο και σε επίπεδο ανθρωπιστικό ιδιαίτερο στο άμεσο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να είχαμε μια ηλεκτρονική επικοινωνία από πλευρά του Επιτρόπου, να μας ενημερώνει δηλαδή τα μέλη της Επιτροπής μας ε, απευθείας μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να γνωρίζουμε τι συμβαίνει και να μπορούμε και εμείς να ενημερώνουμε με τη σειρά μας αλλά εν να διατηρείται και η κινητικότητα στην υπόθεση αυτή. Και επίσης όταν πολύ συχνά ακούγονται επικρίσει γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προχωρεί σε ταχύ ανάληψη δράση κτλ. Και μετά υποβάλλονται αυτέ ή διαβιβάζονται αυτέ οι ε, κατηγορίε είτε στην ύπατη εκπρόσωπο είτε σε έναν επίτροπο, βλέπουμε ότι όντω είχε αναλυφθεί δράση, αλλά δεν ήμασταν ενήμεροι. Γι' αυτό καλό θα είναι να είμαστε ενήμεροι για να ε, διαβιβάζουμε, όπω λέω, τη σχετική ενημέρωση και στα κράτη-μέλη. Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι είτε πρόκειται για την Τρίπολη, είτε πρόκειται για κάποια άλλη πόλη της Λιβύης, διαπιστώνεται μεγάλο χάο στα αεροδρόμια. Ο κόσμος συνοστίζεται, περιμένει ουρά, ε, του δίνουν εισιτήρια για να φύγει με κάποιο αεροπλάνο που τελικά δεν απογειώνεται. Πολλές πιέσεις ε, και ξέρουμε ότι και οι δικοί μας ε, οι πολίτες αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες εκεί. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει δυνατότητα από πλευρά τη ανθρωπιστική ε, τη για τα ανθρωπιστικά θέματα υπηρεσία Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει αυτού του ανθρώπου, έστω πολύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να έχουν μια ανθρώπινη αντιμετώπιση. Γιατί τελικά αυτό που συμβαίνει κατά πάσα πιθανότητα είναι ότι, κάποια, ε, ε, ότι τα φαινόμενα αυτά οφείλονται στην διαφθορά που επικρατεί και σε κάποιου διεφθαρμένου υπαλλήλου εκεί πέρα που προσπαθούν να πάρουν πίσω λεφτά. Κύριε Μπέρμον. Ευχαριστώ την Επιτροπή. Ήταν πολύ συγκεκριμένα τα όσα μας είπε. Πολύ ενδιαφέροντα. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν εάν θεωρεί η Επιτροπή ότι οι προσπάθειες που καταβάλουν τα κράτη-μέλη επαρκούν και αν πιστεύει ότι ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών και των υπηρεσιών της Επιτροπής είναι επαρκής. Κύριο Σφένσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τώρα έχει προκύψει το μεγάλο ζήτημα το τι θα συμβεί εάν αποφασίσει ο Καντάφη όντως να στρέψει το βαρύ του πυροβολικό, τα όπλα του κατά των πολιτών και δει από αέρας. Άνθρωποι όπως εγώ ή φαντάζομαι και οι λοιποί συνάδελφοι που ενδεχομένως δεν έχουν τόση πολύ γνώση της υπόθεσης ε, ε, ε, διερωτώμεθα τι μπορεί να συμβεί, τι έκβαση μπορεί να έχει αυτή η υπόθεση και σε επίπεδο προσφύγων, γιατί θα έχουμε διαστάσεις ρευμάτων προσφυγικών άνευ προηγουμένου. Βλέπουμε διαρκώς κάποιες ειδήσει για πρόσφυγες ε, σε κατάσταση απόγνωσης, είτε πρόκειται για τον Μπαγκλαντές, είτε πρόκειται για οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου, βλέπουμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Αλλά είναι μακριά μας Και τώρα ξαφνικά βλέπουμε από την άλλη όχθη της Μεσογείου ότι είναι δύσκολο ακόμα και να μεταφέρουμε τους δικούς μας πολίτες με τα αεροπλάνα σε ένα ασφαλέ μέρος Ή να βρούμε κουβέρτε να του ε, να τους προσφέρουμε. Νομίζω ότι αυτά είναι απλά πράγματα. Όταν άρχισαν να κλειδονίζονται η Τινησία και η Αίγυπτος ε, αντιλήφθημε ότι θα ακολουθήσει και η σειρά της ε, Λιβύης και ότι τα πράγματα εκεί θα είναι πολύ χειρότερα. Γιατί όταν μιλάμε για τον Καντάφη, ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι ένα άνθρωπος με τον οποίο δεν μπορούμε να έχουμε καμία ε, ε, συνεννόηση. Και γι' αυτό είχαμε πει ότι θα πρέπει να αποσταλούν αντιπροσωπείες, θα πρέπει να αποσταλούν ομάδες γιατρών, να βοηθήσουμε. Όλα αυτά πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ όμω ο κόσμο υποφέρει και χρειάζεται να αναλυφθεί δράση σε διεθνές επίπεδο ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ κύριος Νόησα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που θέσατε και τόσο, τόσο σύντομο διάστημα το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Είναι σημαντικό. Από αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνουν ότι από τις 23 Φεβρουαρίου είναι έτοιμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήδη δύο εβδομάδες δηλαδή. Και ήταν σαφές ότι θα έχουμε ρεύμα προσφύγων προς ε, την Ισία και προς Αίγυπτο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ε, εργαζόμενοι στην Λιβύη, κυρίως από την Αίγυπτο. Η κατάσταση που εμφανίζεται τώρα δείχνει καθαρά ότι δεν επαρκούν οι δυνάμεις του Τινησιακού στρατού για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. Χιλιάδες προσπαθούν να περάσουν και κυρίως Αιγύπτιοι. Εδώ απαιτείται να αναλάβει δράση και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες μέλη. Να προσφέρουν δηλαδή τα τεχνικά μέσα για να μπορούν να φύγουν οι άνθρωποι αυτοί. Κάθε ένας που θα μπορέσει να ε, μεταφερθεί στην πατρίδα του, για παράδειγμα στην Αίγυπτο, θα βοηθήσει να μειωθεί η ένταση. Εμείς μπορούμε να προσφέρουμε την τεχνική αυτή υποστήριξη. Δεν κατανοώ πώς είναι δυνατόν οι χώρες μέλη να κάνουν τόσο λίγα πράγματα. Άκουσα σήμερα το πρωί, για παράδειγμα, από το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, ότι ήρε τώρα την σύσταση μη Μετάβαση τουριστών στην Αίγυπτο. Άρα δηλαδή τώρα μπορούν να πάνε οι Γερμανοί τουρίστες στην Αίγυπτο και παρόλα αυτά δεν καταφέρνουμε να προσφέρουμε επαρκή τεχνική υποστήριξη για να μεταφερθούν οι άνθρωποι από την παραμεθόριο περιοχή Λιβύης στην Ισίας προς την Αίγυπτο. Η κατάσταση αυτή μπορεί να επιδεινωθεί ανα πάσα στιγμή. Εάν κλιμακωθεί ο εμφύλιος, η εμφύλια σύραξη ανάμεσα στο δυτικό και το ανατολικό μέρος της ε, Λιβύης. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν πολύ περισσότερα και ως Ένωση και ως χώρες μέλη. Έχει το λόγο κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις. Τι ακριβώς κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει την, την Ισία να υποδεχθεί αυτούς τους πρόσφυγες Είπατε τα χρήματα, αναφέρατε τα ποσά που θα δοθούν, αλλά για ποιο λόγο ακριβώς. Τα προγράμματα επαναπατρισμού δεν θα εξυπηρετήσουν όλους τους πρόσφυγες που βρίσκονται τώρα στην Τινησία. Δεύτερο, έχει γίνει τίποτα για τους πρόσφυγες από Σομαλία και Ερυθρέα τους οποίους ξαναστέλνει στη Λιβύη η Ιταλία επομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση και πού πάνε αυτοί οι άνθρωποι, σε στρατόπεδα στη Λιβύη, στην έρημο. Τι γνωρίζουμε για την κατάστασή τους. Κυρία Θεοχάρου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι η βοήθεια που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η Λιβύη και οι χώρες κοντά στη Λιβύη δεν είναι αναπτυξιακή βοήθεια. Είναι βοήθεια άμεσης παρέμβασης για να διασωθούν οι άνθρωποι. Οι οποίοι μέσα σε κλίμα πανικού κυρίως τρέχουν να φύγουν από τον εμφύλιο. Δυστυχώς ποτέ δεν έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά για να ακούμε τα μηνύματα των καιρών. Και να σας θυμίσω ένα παράδειγμα τους Χούτου και τους Τούτσι στην Ρουάντα που ξέραμε ότι θα γίνει. Αυτή τη στιγμή αναρωτιόμαστε αν θα κάνει εγκλήματα αυτός ο αιμοσταγής δικτάτορας ο Καντάφη. Να θυμίσω ακόμη ότι σε άλλες περιπτώσεις όπως στη Γάζα οι άνθρωποι δεν μπορούν να φύγουν γιατί τα σύνορα είναι μονίμως κλειστά. Άρα το σκηνικό στην Βόρεια Αφρική είναι τέτοιο που να επιβάλλει εκείνο που έχει πει και η κυρία Σίρφλερ στην έκθεση της και άλλες φορές έχουμε πει για την, δημιουργία, την ανάγκη δημιουργία μιας ομάδας άμεσης παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτά που συμβαίνουν τώρα. Επιχείρησα να μεταβώ στη Βενγάζη ως χειρουργός την περασμένη εβδομάδα, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό Θέλω να σας πω ότι η υποδομή στην Βόρειο Αφρική, στην Λιβύη ειδικά, είναι πάρα πολύ καλή. Δεν χρειάζονται αυτή τη στιγμή το νοσοκομεία να τους φτιάξουμε, επαρκούν τα νοσοκομεία. Εκείνο που χρειάζεται είναι να πάνε οι άνθρωποι που μπορούν να τους βοηθήσουν, να πάρουν το υλικό. Και τώρα, όσον αφορά την ανθρωπιστική κρίση των Ευρωπαίων πολιτών ή των ξένων πολιτών, ναι, είναι ένα άλλο ζήτημα που θα πρέπει να γίνεται σε επίπεδο κυβερνητικών και ε, ε, ε, ε λήψης αποφάσεων αλλά όσον αφορά την ροή των προσφύγων για τους ντόπιου τραυματίες και θύματα του πολέμου, ε, ναι, εκεί θα πρέπει να το δούμε μέσα από ένα οργανωμένο μόνιμο σύστημα παρέμβασης. Ε, θα μπορούσα να έλεγα πάρα πολλά αυτά για την ώρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Στίφλερ. Oui, merci beaucoup, Madame euh, la Présidente. Je rejoins tout à fait ce que dit Madame. Δέχομαι απόλυτα αυτά που είπε η κυρία Θεοχαρού. Σας μη συγχαίουμε ανθρωπιστική βοήθεια και αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτό που με απασχολεί είναι οι 40.000 άνθρωποι που είχαν αποκλειστεί στα σύνορα και έχουν εξαφανιστεί. Θα πρέπει να είμαστε ε, δυστυχώς σε μια κατάσταση ε, άμεσης αντίδρασης, διότι με τον Καντάφη οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Και όπως είπε ο κύριος Μίτσελ, θα πρέπει να παρακολουθούμε την κατάσταση εν τη εξελίξη της γιατί ανάλογα ο τύπος ανάλογα με τη διάθεση των δημοσιογράφων μπορεί να μας δώσει ανακριβή στοιχεία. Γι' αυτό θα ήθελα να έχουμε πληροφορίες κατά τη διάρκεια, κατά την εξελικτική πορεία των γεγονότων. Ο κύριος Ντέβα, ευχαριστώ πρόεδρε. Υπάρχουν ε, δύο τρόποι σκέψης που απορρέουν από τη συζήτηση. Αφενός, δεν μπορούμε να προτρέξουμε ως προς τις ε, κρίσεις αυτές που ανακύπτουν ως προς θέματα χρονισμού και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το χειρότερο. Γιατί δεν μπορούμε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας παρά σε καταστάσεις παρά μόνο όταν έχουν επισυμβεί. Θα πρέπει να μπορούμε να προτρέξουμε λοιπόν και να δράσουμε εντάχει. Το δεύτερο θέμα έχει ως εξής. Έχοντας αντιδράσει βέβαια, η Κομισιόν δεν μπορεί να ερμηνεύσει τα γεγονότα. Εγώ πολλές φορές ε, ρώτησα τι κάνει η Κομισιόν γιατί δεν το βλέπουμε στα νέα, ούτε στο Euronews, ούτε στο CNN. Και φαίνεται σαν να έχουν αποχωρήσει, σαν να κάνουν διακοπές, κάτι το οποίο δεν ευσταθεί, αλλά υπάρχει, επικρατεί αυτή η αντίληψη. Άρα μου τηλεφωνούν εμένα ή τον κύριο Μίτσελ και μου λένε «Μα τι κάνει επιτέλους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στον τύπο. Γιατί μέσω blog, Twitter, SMS και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά, όλες αυτές τις τεχνολογίες εχμής, γιατί να μην τις χρησιμοποιούμε. Όταν ε, ε, δεν, όταν θα μπορούσαμε να αντιδράσουμε άμεσα, να ξέρουμε πώς έχει η κατάσταση και να μην τα γράφουμε δύο εβδομάδε μετά, να μην γράφονται επί χάρτου δύο εβδομάδε μετά. Θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή τι μπορεί να κάνει για τους πολίτες της, ε, του Νοτίου Σαχέλ που, γιατί εδώ υπάρχει μία σύγχυση με τους Λίβιους και τους μισθοφόρους του Καντάφη. Από την άλλη πλευρά θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο η Frontex έχει οδηγίες έτσι ώστε οι πρόσφυγες να μεταφέρονται ε, από εκεί που, εκεί, από όπου προέρχονται ή θα πρέπει να έρχονται προς τα εμάς. Υπάρχει το καθεστώς του προσωρινού πρόσφυγα του 2001 ισχύει και νομίζω ότι τα ποσά που προβλέπονται σήμερα, 3 εκατομμύρια δηλαδή ευρώ και 17 εκατομμύρια ευρώ για την Τινησία, είναι εντελώς ανεπαρκή. Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την έκριθμη κατάσταση και δεν μας τιμούν. Δεν θα πρέπει να αυξήσουμε την επιμελητιακή βοήθεια και τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Η κυρία Τζίμερ. Εγώ παρακολούθησα προσεκτικά την συζήτηση όπως διεξήχθη μέχρι τώρα. Συμφωνώ με πολλές από τις ερωτήσεις που έκαναν άλλοι συνάδελφοι. Μου φαίνεται όμως σημαντικό και το εξής ερώτημα απευθείας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μήπως είναι τόσο δύσκολο να συμφωνήσουν πάνω σε μια νέα στρατηγική άμεσης βοήθειας επειδή μέχρι τώρα η στρατηγική απέναντι στη Λιβύη ήταν τελείως διαφορετική επειδή κυρίως ασχολούνταν να δουν πώς μπορούν με τη βοήθεια της Λιβύης να ανακόψουν τα μεταναστευτικά ρεύματα προς την Ευρώπη. Και τώρα έχουμε δυσκολία να αντιληφθούμε ότι η στρατηγική αυτή ήταν απολύτως εσφαλμένη, οδήγησε στο μηδέν και εμφανίζεται σήμερα να είναι καταστροφική. Τι κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε τώρα σε αυτή την κατάσταση να αλλάξει απολύτως πορεία. Από το 2008 είχαμε επισημάνει την παγκόσμια κρίση πείνας και τότε είχε εξασφαλιστεί να κονδύλι ενό δισεκατομμυρίου για να αντιδράσει. Ακούσαμε πριν ορισμένα ποσά τα οποία υποτίθεται θα διατεθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσαμε και τα λεφτά που δίνουν οι χώρες μέλη είναι ντροπιαστικά τα ποσά αυτά, παραπάνω από ντροπιαστικά. Αυτό το σχόλιο το απευθύνω σε εσά, αλλά το απευθύνω βεβαίω και στι χώρε μέλη. Όταν η Γερμανία εμφανίζεται με 660.000 ευρώ, πρόκειται στην ουσία για μια, ένα πραγματικό έσχο. Πάντω, θα ήθελα να μου, κάνει, να μου δώσετε ξεκάθαρε απαντήσει στα δύο τουλάχιστον πρώτα ερωτήματα. Donc, euh, monsieur le... Ευχαριστώ. Κύριε εκπρόσωπο της Επιτροπής, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ίσως παρέμουν συνοπτικό στην παρουσίασή μου, αλλά θα προσπαθήσω να δώσω απαντήσεις στην κάθε ερώτηση. Οτιδήποτε δεν μπορώ να απαντήσω τώρα, πολύ ευχαρίστως να ερευνήσω, Πρόεδρε, και πρόκειται για την ερώτηση της, για τη Frontex συγκεκριμένα για την οποία δεν έχω πληροφορίες ε, τελευταίες στο θέμα αυτό. Για το κατά πόσον υπάρχει επίσημο συνομιλητή σε επίπεδο αρχών Λιβύης. Για να σε αυτά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μεταβούμε, δεν μπορούμε να μπούμε στην Τρίπολη. Είναι υψηλότατος, ο υψίστος ο κίνδυνος, ε, δεν μπορούμε να στείλουμε ειδικό, ούτε δικό μας, ούτε από αραβική χώρα. Και ως εκ τούτου, για τη δική μας την DG, τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ, δεν υπάρχει συνομιλητής επίσημος από πλευράς Λιβύας. Προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε θεώρηση διαβατήριο στην αρχή της κρίσης από την ε, πρεσβεία της Λιβύης στο Αμάν της Ιορδανίας. Αλλά όταν ήρθε η ώρα να παραλάβουμε τις, ε, να πάρουμε την απάντηση, μάθαμε ότι ο πρεσβευτής είχε παραιτηθεί, δεν υπήρχε τρόπος να μεταβούμε, να μπούμε στην ε, Λιβύη. Επίσημώ, Ο μόνος λοιπόν συνομιλητή αυτή τη στιγμή είναι ο Ερυθρός Σταυρός, λέει ο μιλητή. Για την χρηματοδότηση υπάρχουν δύο συγκρουόμενες απόψεις. Ότι πολλά γίνονται αφενός, ότι δεν γίνονται αρκετά αφετέρου. Για την Επιτροπή μπορώ να πω το εξής. Ο πρόεδρος είπε ξεκάθαρο ότι χρειάζονται περισσότερα πράγματα να γίνουν. Σε αυτό το θα εμεί και έτσι προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε περισσότερα κονδύλια. Αλλά αυτό θα γίνει σε στάδια. Στην απαρχή μια κρίση και όταν δεν γνωρίζουμε τι πρόκειται να συμβεί συγκεκριμένα, δεν μπορεί να πει κανεί θα ρίξω 50 εκατομμύρια ευρώ όταν το πρόβλημα δεν έχει προσδιοριστεί επαρκώ. Χρήματα υπάρχουν, είναι διαθέσιμα. Το ξέρουν και οι οργανώσει μα ότι είναι διαθέσιμα τα κονδύλια και πριν ακόμη να εμφανιστούν πρόσφυγες στα σύνορα της Τινησίας είχαμε τους, ε, την κυρία Τζεωτζίεβα και τους άλλους αδέλφους που λέγανε, εξηγούσαν τι πρόκειται να γίνει και τι μπορούμε να προσφέρουμε. Είναι σε υψηλό βέβαια επίπεδο επικαιρότητας για μας η Λιβύη, αλλά εξίσου και για την Επίτροπο Γεωργίευα και για εμά όλου έχει σημασία η αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Που μπορεί να μετατραπεί σε φίλιο πόλεμο και να ε, αποσταθεροποιήσει και άλλα γειτονικά κράτη όπω τη Λιβυρία. Λιβερία. Άρα λοιπόν παρακολουθούμε την κατάσταση και θα λάβουμε όταν έρθει η ώρα την κατάλληλη απόφαση. Πάντω προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι στο βαθμό του δυνατό. Επίση η Επίτροπο Γεωργίευα ε, προσπαθεί να ενισχύσει τη χρηματοδότηση για την ε, πιο λησμονημένη κρίση, τη Σαλχάουι δηλαδή, αλλά και για την Ιεμένη. Δεύτερον, μέγιστο μέλημά μας, έψιστο μέλημά μας αυτή τη στιγμή, η περιοχή μέσα στη Λιβύη που βρίσκεται σε επίπεδο κάτω από τη Σαχάρα όπου υπάρχουν άνθρωποι ε, που έχουν πάει να κρυφτούν, φοβούνται μην τους ε, πάρουν για μισθοφόρους και τους φωνεύσουν. Αυτό είναι το μεγάλο μας μέλημα αυτή τη στιγμή για την ίδια τη Λιβύη και ιδιαίτερα της, ε, και δικό μας μέλημα και της ΥΠΑ της Αρμοστίας. Και έτσι και με την Εθνή Οργάνωση Μεταναστών και με την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία προχωρούμε σε συντονισμό ε, των προσπαθειών μας ώστε να στηρίξουμε κάθε έναν που πλήττεται από αυτή την ε, σύγκρουση στη Λιβύη. Όχι, δεν κοιτάμε δηλαδή που θα πάνε τα χρήματα, θα πάνε στη Λιβύη, την ε, Αίγυπτο, την Τινησία. Κοιτάμε, όπως είπα, και τον Ήγυρα και τα Αλγερινά σύνορα. Στον Ήγυρα έχουμε μέσο διαμετακόμισης. Οι υποσαχάριοι πληθυσμοί δηλαδή καλύπτονται και από την ανάλυση μας. Αλλά και από τη χρηματοδότηση. Ροή πληροφοριών λυπούμε που θεωρείτε πως δεν ενημερώνεστε επαρκώς. Εμείς κάθε μέρα, κάθε βράδυ συγκεκριμένα αποστέλουμε ενημέρωση με την έκθεση επικαιρότητα στη γραμματεία. Φαίνεται ότι δεν λειτουργεί αυτό ο τρόπος επικοινωνίας, θα το συζητήσουμε και πάλι. Πάντω, εμείς κάθε μέρα στέλνουμε τις πιο ε, πρόσφατες πληροφορίες που έχουμε στη θέση μας για να είναι ενήμερα τα μέλη της Επιτροπής σας δεν υπήρχε καμία πρόθεση από πλευρά μα να μην σα ενημερώσουμε τον αντίον μάλλον. Θα το συστήσουμε απευθεία με τη γραμματεία και ελπίζω ήδη σήμερα το βράδυ να έχετε την έκθεση επικαιρότητα. Κάθε μέρα και χωρίς καθυστέρηση. για τις ε, αντιπροσωπείες. Δεν έχουμε αντιπροσωπεία στην Τρίπολη πρώτον και δεύτερον ε, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν ήταν και τόσο ευπρόσδεκτε στα τελευταία χρόνια στη Λιβύη. Ως εκ τούτου είπατε αρμοστία ε, λίγο πολύ ε, βρέθηκε έξω από την πόρτα μας το 2010 ε, έχουν 2.500 περίπου ανθρώπου σε ένα κατάλογο αναμονή, έχουν του πρόσφυγε με του οποίου προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά του και δεν φτάνουν αυτά. Ξέρουμε ότι υπάρχουν 25.000 Παλαιστίνοι στη Λιβύη, εκ των οποίων 23.000 δεν έχουν κανένα νομικό καθεστώ Ωστόσο αυτό έχουμε να κάνουμε μια χώρα στην οποία ούτως ή άλλω ήταν δύσκολη η δουλειά των ανθρωπιστικών οργανώσεων. Και είναι δύσκολο να λάβουν τώρα δράση το ανθρωπιστικό προσωπικό τώρα, αυτό που βρίσκεται στην Τρίπολη, είναι ε, βρίσκεται κρυμμένο, δεν κυκλοφορούν ανοιχτά γιατί φοβούνται και για τη δική τους την ασφάλεια. Υπάρχει συντονισμός βέβαια, εν εξελίξη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση χάρη στην Ουγγρική Πρεσβεία που παραμένει με το προσωπικό της και οργανώνει το συντονισμό καθημερινά για τη βοήθεια. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να προσφερθεί βοήθεια και πρέπει να πω επίσης ότι ναι, έχουμε καλό συντονισμό. Ο, η συγχώνευση μεταξύ του δυναμικού πολιτικής προστασίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας νομίζω λειτουργεί. 8.30 κάθε πρωί έχουμε συνάντηση και μερικές φορές ακόμη και το βράδυ, δεύτερο συντονισμό. Το Κέντρο Παρακολούθησης και Πληροφοριών συντονίζει τις προσπαθίες του με τα κράτη-μέλη Περίπου 80.000 είναι οι άνθρωποι που έχουν περάσει από την Αίγυπτο και από την εκεί πλευρά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Περίπου ο ίδιος αριθμός προσφύγων που έχουν μεταβεί από την άλλη πλευρά προς την Τινησία αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η Το δυναμικό μα ενισχύεται διαρκώ και περιμένουμε από τα κράτη-μέλη μέχρι σήμερα το 12 το μεσημέρι να μα πούν εάν είναι διατεθειμένα να προσφέρουν επιμελητιακή υποστήριξη, μέσα υποστήριξη για άμεσο επαναπατρισμό αυτών των πολιτών. Και θα δούμε ποια είναι η απάντηση. Το Ρημένο Βασίλειο και η Γαλλία, όπω είπα, ήδη έχουν αναλάβει δράση. Το Εξωτερικών της Ιταλίας, ο Υπουργό Εξωτερικών τη Ιταλία επίση δήλωσε ότι πρόκειται να προσφέρει την επιμελητιακή βοήθεια που χρειάζονται οι πολίτε τη χώρα του. Τη μεταφορά. Ο συντονισμός με τα κράτη-μέλη λειτουργεί πολύ καλά. Έχει λειτουργήσει καλά η εκένωση Ευρωπαίων ε, υπηκών. Τώρα πρέπει να δούμε με την Τινησία πώς μπορούμε να βγούμε από, το, από τις θενοπούς και να πείσουμε τις τινησιακές αρχές να ανοίξουν τα σύνορα. γιατί ε, η περιοχή αυτή φαίνεται να, έχει, να γνωρίζει πολλές ε, πιέσεις μεταναστευτικές ή προσφύγων. Για τη Σομαλία και την Ερυθρέα βεβαίως θα προσφέρουμε την υποστήριξή μας και για, την, ε, για τον επαναπατρισμό και για την άμεση βοήθεια. Έχουμε και πολλούς Παγκλαντέσιανούς που χρειάζονται βοήθεια. Επιμελητιακά έχουμε το πρόβλημα ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους έχουν αφήσει τα διαβατήριά τους έχουν φύγει από τη χώρα, φτάνουν στην Αίγυπτο και δεν έχουν ε, τρόπο, δεν έχουν προσωπικά έγγραφα για να ε, αναγνωριστούν επικότητα κτλ. Και εμεί προσπαθούμε να τους πείσουμε, να τους βοηθήσουμε πριν να τους ε, προωθήσουν προς άλλο αεροδρόμιο οι αρχές της Αιγύπτου ή πριν αποχωρήσουν από τη χώρα. Όπως είπα, αυτέ οι 40.000 είναι ανησυχητικό είναι λόγος φυσικά, δεν μπορεί κανείς να περάσει τα σύνορα νησία Λιβύης. Έχουμε τι οργανώσεις μας, έχουμε την Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού, έχουμε κάνει έκκληση για ανθρωπιστική πρόσβαση, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει δυνατότητα να μπούμε από τα σύνορα της Τινησίας στη Λιβύη, δηλαδή στο δυτικό τμήμα της χώρας το πώ θα μπορούμε να προβλέψουμε ή να, προλάβουμε μια κρίση. Ναι, όντω μπορούσαμε να προβλέψουμε ότι κάτι θα γίνει. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετέ χώρε στην περιοχή όπου αναπτύσσονται διαδηλώσει, συλλαλητήρια, τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν πάρα πολύ γρήγορα. Ε, φυσικά παρακολουθούμε στενά τι εξελίξει αυτέ και παρόλα αυτά θα ήταν ε, μη σόφρον αυτή τη στιγμή να δηλώσουμε ανησυχία δημόσια σήμερα για τις εξελίξεις και να εξηγήσουμε ότι σκοπεύουμε να οργανώσουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Γιατί αυτό τελικά μπορεί να οδηγήσει στην πρόκληση του προβλήματος. Πάντως οργανώνουμε όσο μπορούμε τις, ε, ε, το δυναμικό μας και κυρίως από πλευράς Τινησίας και Αιγύπτου βελτιώνουμε την παρουσία μας εκεί και ζητούμε από τους ειδικού μας να μας ενημερώσουν καθημερινά, όπως μας ενημερώνουν βέβαια και οι αντιπροσωπείες ε, της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και τα κράτη-μέλη. Για τη χρηματοδότηση, και μια και ακούστηκε και η Γερμανία. Πιστεύω ότι θα πρέπει τώρα να αντιληφθούμε ότι εάν ε, μέσα σε δύο μήνε δεν προσφερθούν περισσότερα κονδύλια, ναι, μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Αλλά αυτή τη στιγμή το πρόβλημα δεν είναι χρηματοδότηση. Έχω λάβει ήδη δεσμεύσει οικονομικέ από την Επιτροπή, ένα εκατομμύριο από τι ΗΠΑ, 500.000 ελβετικά από του Ελβετού. Το πρόβλημα δεν είναι λοιπόν το οικονομικό. Το πρόβλημα είναι να βρεθούν τα σκάφη και τα αεροσκάφη, η επιμελητία και ο συντονισμό που χρειάζεται να ε, ξεκινήσουν και να λειτουργήσουν ώστε να φύγει ο κόσμο από εκεί μέσα. Η Επίτροπο Γεωργίευμα, όπω είπα, μάλλον θα ενισχύσει, θα ε, προσφέρει περισσότερα κονδύλια από αυτά που ήδη είναι διαθέσιμα και τα κράτη-μέλη νομίζω ήδη έχουν μπει σε αυτήν την τροχιά. Έχουμε πληροφορίες ε, ικανοποιητικές για την πλευρά της Τινησίας, έχουμε καλές πληροφορίες για τόσα συμβαίνουν στην Μπενγκάζη και πρέπει να πω ότι η Βενγκάζη δεν έχει πρόβλημα ανθρωπιστικό αυτή τη στιγμή. Ορισμένα φάρμακα λείπουν, αλλά το κυριότερο πρόβλημα στο, για το φαρμακευτικό σύστημα είναι η απουσία προσωπικού, γιατί έχουν φύγει οι γιατροί και νοσοκόμοι. Στη Βεγγάζη λοιπόν πιο πολύ μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή η κατάρτιση και όχι η λειτουργία, όχι η δράση. Είναι ήρεμη η κατάσταση. Όπως είπα μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξει και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Αυτό που μας ανησυχεί είναι η μαύρη τρύπα, 100 χιλιόμετρα νότια της Βεγγάζης, όπου δεν έχουμε πρόσβαση ούτε στην περιοχή της Τρίπολης, ούτε γύρω από την Τρίπολη ε, και όπου φοβούμαστε, ιδιαίτερα για τους υποσαχάριους Αφρικανούς, ότι εκεί ακριβώς θα εντοπιστεί το πραγματικό ανθρωπιστικό πρόβλημα πέραν των όσων έχουμε στα σύνορα της Τινησίας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε λοιπόν για να συλλέξουμε στοιχεία. Ζητούμε και από τους ειδικού μας να προσπαθήσουν να δούνε ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες προοπτικές όσον αφορά την προμήθεια σε τρόφιμα, ώστε εάν υπάρξει κίνδυνο σε τρεις-τέσσερις εβδομάδες να, να εμφανιστεί παινία η σπάνιδα τροφίμων, να έχουμε τη δυνατότητα να φέρουμε προς το τρόφιμα στη χώρα. Ελπίζω να έδωσα απαντήσεις τουλάχιστον στις περισσότερες ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Οπωσδήποτε θα τα ξαναπούμε για αυτό το θέμα. Περνάμε τώρα στο θέμα 7 της ημερήσιας διάταξης. Εντάχει, εντάχει. Ζητώ συγγνώμη, Φτάσα αργά γιατί καθυστέρησε το αεροπλάνο. Θα ήθελα να σας πω ότι η Ιταλία έχει αναλάβει ενεργό δράση. Ίσως ξεχνάτε ότι εδώ και μήνες η Ιταλία ζητά βοήθεια από την Ευρώπη και από όλα τα κράτη-μέλη. Μην ξεχνάμε ότι φτάνουν αυτοσχέδια πλοία με... και φτάσανε χτες 400 άνθρωποι που βρίσκονται σε ικτρή κατάσταση και πρέπει να υποστηρίξουμε 10.000 ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτάσει. Μην ξεχνάτε ότι ο Υπουργός Μαρών ήταν εδώ και σας ζήτησε βοήθεια. Μην ξεχνάμε ότι στην ουσία αντιδρούμε πολύ αργά. Εδώ και μήνες ζητά η Ιταλία βοήθεια από την Ευρώπη και ε, η Ευρώπη δεν αντιδρά καν. Πρόκειται για, βοή, ε, για φωνή βόντος εν τη ερήμο. Χρειαζόμαστε βοήθεια γιατί πρόκειται για ανθρώπους που βρίσκονται σε κατάσταση απόγνωσης. Μην ξεχνάτε ότι ούτε η Λαμπετούσα ούτε η Παντελερία τα βγάζουν πλέον πέρα. Μιλάμε για 10.000 πρόσφυγες που φτάσουν και βρίσκονται σε ικτρή κατάσταση. Πρέπει να μας βοηθήσετε, Πρόεδρος. Τώρα θα ασχοληθούμε με τις ψηφοφορίες. Επειδή υπάρχουν πολλές ψηφοφορίες, θα κάνουμε μία δοκιμή καταρχήν. Σας παρακαλώ βγάλτε τις κάρτες σας. Χέλλερ, υπάρχει ένα τεχνικό θέμα, διότι υπάρχει η τροπολογία 2 του κυρίου Ντέβα για τις μεταναστευτικές ροές, όπου υπάρχουν δύο διαφορετικά αριθμητικά στοιχεία. Φαίνεται ότι και τα δύο είναι σωστά. Αυτά τα στοιχεία που βασίζονται θα πρέπει να το γνωρίζουμε πριν ψηφίσουμε. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν πληροφορίες επί του θέματος. would Mrs. Keller be a little bit more specific? Are you questioning... Τι αμφισβητείτε? Το ένα δις... Ποια, ποιο αριθμητικό στοιχείο, για ποιο αριθμητικό στοιχείο μιλάτε, ποιο αμφισβητείτε. Hm? The failed state index says that after... Γίνεται λόγος για 38 ευάλωτα κράτη. Και η Παγκόσμια Τράπεζα λέει ότι πλήττονται, πλήττεται ένα δισεκατομμύριο από αυτή την κατάσταση. Εσείς ποιο αριθμητικό στοιχείο αμφισβητείτε. Κάποιοι άλλοι μίλησαν για 34 και 600 εκατομμύρια που πλήττονται από αυτή την έκρηθμη κατάσταση. Και η συντάκτρια δεν είναι εδώ για να μας πει από πού προέρχονται τα αριθμητικά στοιχεία που μας δίνει. Δεν ξέρω αν ξέρει κάποιος Έχει τόση σημασία αν μιλάμε για 34 ή 38 ευάλωτα κράτη. Έχει τόση μεγάλη σημασία. Ε, μιλάμε για τρόπο υπολογισμού, δηλαδή εδώ πρόκειται για τρόπο υπολογισμού δεν είναι θέμα ουσίας. Θα επαληθεύσουμε αυτό το, αυτά τα στοιχεία εάν εγκριθεί η τροπολογία. Ωραία, να κάνουμε μια δοκιμή. Με τις κάρτες αρχίζει η ψηφοφορία. Βάλτε κάρτες παρακαλώ. Δοκιμή, δοκιμή απλώς. Ένας ή μία δεν ψήφισαν. Ίσως εγώ, λέει η πρόεδρος, εγώ ήμουν αυτή. Εγώ δεν είχα ψηφίσει. Μπορούμε να αρχίσουμε λοιπόν. Θα ψηφίσουμε Ε, διανατάσεως της χειρός την έκθεση της Κορίνα Κρέτσου για τη μετανάστευση. Τροπολογία Ντέβα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Στη συνέχεια. Τροπολογία 1, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ, Με συγχωρείτε, λέει η Με συγχωρείτε, πέντε Υπέρ. Υπέρ τις πέντε Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία έξι Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία επτά Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 11. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτω. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός α υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 17 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία, προφορική τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές θα πρέπει να επαληθεύσουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός Β υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να επαληθεύσουμε επί του συμβιβασμού Β. Ωραία, αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Adopté, donc... Oral Amendement oral. Προφορική 2. Ε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 31. Όχι, όχι. 31, 31 υπέρ. Κατά αποχές καλύτερα να επαληθεύσουμε αρχίζει η ψηφοφορία επί της 31 ψηφίσατε όλοι πέρασε εγκρίνεται 32. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές. Καλύτερα να ελέγξουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε την γνωμοδότηση όπως έχει τροποποιηθεί ηλεκτρονική ψηφοφορία η οποία και αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Voilà.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 ένα έχει αποσυρθεί, δύο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την γνωμοδότηση στο σύνολό της ηλεκτρονικά πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται ομόφωνα. Στη συνέχεια ψηφίσουμε την έκθεση DEVA. Μπορούμε να ψηφίσουμε unblock. Έκθεση ΔΕΒΑ, έκθεση για θέματα αλίας, αλλιευτικής σύμπραξης, μπλοκ υπέρ όλων των τροπολογιών κατά αποχές εγκρίνονται. Άρα εγκρίνεται ομόφωνα. Θέλετε να παληθεύσουμε, ωραία, ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Χωρίς καμία έκπληξη ομόφωνα λοιπόν. Τώρα θα ψηφίσουμε την έκθεση Σνίπερ Γιάστραν, Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, έχει απορριφθεί η πρώτη. Ωραία, ωραία. Ας επαληθεύσουμε. 5. Έλεγχος. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβασμός 2 υπέρ. Α, έχουμε ξεχωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10. Τροπολογία υπαριθμών 10. Ξεχωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σημειώσμος 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 τμήματική ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Α, καταπίπτει. 16 λοιπόν, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19. Τμηματική και πάλι. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προφορική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 τμηματική και πάλι πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Ας ελέγξουμε καλύτερα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20 ή 23 καταπίπτει, λέει πρόεδρος. 25, 25 λοιπόν. Περνάμε στην 25, αρχίζει η ψηφοφορία. Μάλλον με συγχωρείτε, λέει πρόεδρος. Έχει απορριφθεί η τροπολογία συμβασμού υπαρτμούν 3, άρα ψηφίζουμε την 25, 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αρχίζει η ψηφορία, λέει η πρόεδρος. Ψηφίσατε όλοι. Πέραστε. Απορρίπτεται. Για μία ψήφο. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Καλύτερα να ελέγξουμε, λέει η Πρόεδρος. Επαληθεύουμε το πρώτο τμήμα της 27. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28. 28 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 ξεχωριστή τμηματική πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε ε, ε, ηλεκτρονικά επί της, ε, του σχεδίου γνωμοδότησης. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν ομόφωνα. Τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες. Bon, en plus, il y avait beaucoup de votes à une voix, quoi.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 Euh, Συνεχίζουμε τη συνεδρίαση. Παρακαλώ να καθίσετε και πάλι. Ευχαριστώ πολύ που καθίσατε και πάλι. Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω τον κύριο Σέικ Σιντιτζιαρά, το εκπρόσωπο για τις λιγότερο ανεπτυγμένε χώρες, τις χώρες χωρίς, ε, που δεν βρέχονται από θάλασσα, και Γενικό Γραμματέα της Διάσκεψης των ΗΠΑ για τις λιγότερο ανεπτυγμένε χώρες, που θα λάβει χώρα, χώρα από τους 9 στις 13 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη που στόχο έχει να αξιολογήσει τη δράση των βρυξελων 2000-2010 για τις λιγότερο ανεπτυχμένες χώρες, ταυτόχρονα όμως θα αποτελέσει και ένα καλό τρόπο να εκτιμηθούν οι βέλτιστες πρακτικές για να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια και να διατυπωθεί μια νέα εταιρική σχέση μεταξύ των λιγότερων ανεπτυγμένων χωρών και των αναπτυσσομένων χωρών εταίρων. Κύριε τινά θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι η Επιτροπή μα απεφάσισε να αποστείλει αντιπροσωπεία στη διάσκεψη αυτή, δεδομένη σημασία που αποδίδουμε στην, στον αγώνα για την καταπλέμιση τη φτώχεια στι χώρε αυτέ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι εθνικοί εταίροι, οι χώρε δηλαδή, έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν προκειμένου να εκδημοκρατιστούν περαιτέρω οι χώρες αυτές και να προχωρήσουν με πολιτικές ανάπτυξης προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα πιο ευάλωτα σημεία που έχουν να κάνουν κυρίως με, την οικονομική κρίση, την ενεργειακή, την ε, επιστηστική κρίση και την κλιματική αλλαγή. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστώ που ήρθατε να μας εξηγήσετε ε, σε μεγάλες ε, αδρές γραμμές τα περί της δίσκεψης Κωνσταντινούπολης. Έχετε το λόγο για 20 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. πολύ ε, καλή είδηση ότι θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τις λιγότερο εμπτυγμένες χώρες. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα η δυνατότητα που μου δίνετε να απευθύνω το λόγο στην Επιτροπή σας για την επερχόμενη τετάρτη διάσκεψη των Αθηνών για τι λιγότερο αναπτυγμένε χώρες, η οποία θα λάβει χώρα στην Κωνσταντινούπολη από τις 9 στις 13 Μαΐου του 2011. Ξεκινώντα, θα ήθελα να σα συγχαρώ για το μεγάλο ενδιαφέρον που δείχνετε προκειμένου να ενημερωθείτε για τι λιγότερο ανεπτυγμένε χώρε και τη βούλη σα να στηρίξετε αυτή τη διαδικασία. Αυτή η στράτευση πιστεύω θα οδηγήσει σε ακόμη ταχύτερε εξέλιξει στις χώρε αυτέ. Όπω γνωρίζετε, οι λιγότερο ανεπτυγμένε χώρε, ω λιγότερο ανεπτυγμένε χώρε, ονομάζουμε τι 48 φτωχότερε και πιο αδύναμες χώρε. Το πιο φτωχό και αδύναμο κομμάτι δηλαδή τη διεθνού κοινότητα. Με χαμηλό κατά κεφάλαιο εισόδημα, πολύ χαμηλή ανάπτυξη του ανθρώπινου του δυναμικού και ιδιαίτερα πολλά σημεία ε, τροτά και ως προς την εσωτερική αλλά και ως προς την εξωτερική τους ε, ανάπτυξη. Αναγνωρίζεται λοιπόν από την διεθνή κοινότητα, από την ΕΕ, η ανάγκη να στηριχθούν τα κράτη αυτά και έχουν θεσπιστεί τρία προγράμματα δράσεω για τι λιγότερο ενδεικμένε χώρε ε, που ξεκίνησε το 1981 στο Παρίσι για να κινητοποιηθεί η παγκόσμια στήριξη για τι κοινωνικο-οικονομικέ εξελίξει τη χώρα αυτέ. Το, το τρίτο πρόγραμμα δράσεω, το λεγόμενο πρόγραμμα των Βρυξελών για τι λιγότερο ανεπτυγμένε χώρε για την περίοδο 2001-2010 Υιοθετήθηκε εδώ, ακριβώς, στις Βρυξέλλες, στην τρίτη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών το 2001. Κύριος και γενικός στόχος αυτού του προγράμματος των Βρυξελών ήταν, παραθέτω, ουσιαστική πρόοδος προς την υποστήριξη, προς την παροχή αρρωγής στους ανθρώπους που ζουν στις περιοχές αυτές και που αντιμετωπίζουν την λιμοκτονία έως το 2015, πέρας παραθέσεως. Δηλαδή, και ενώ προχωρούμε προς τέταρτη διάσκεψη, πιστεύουμε ότι θα έχουμε για ε, τις χώρες αυτές και το πιο αδύναμο κομμάτι του παγκόσμιου πληθυσμού ένα ουσιαστικό πρόγραμμα που θα αποτελεί και αναβάθμιση του προγράμματος των Βρυξελών και την υιοθέτηση ενός νέου προγράμματος για τις, ΛΑΧ, λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, που θα μας οδηγήσει στην δεκαετία 2011-2020. Πριν εστιαστώ στις προετοιμασίες και τις προσδοκίες για την τέταρτη διάσκεψη, επιτρέψτε μου να δώσω μια σύντομη επισκόπηση και αξιολόγηση του προγράμματος των Βρυξελών. Κυρίες και κύριοι, η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, εξέλιξη μάλλον ε, στις λιγότερο εμπτυγμένες χώρες ε, προχώρησε πολύ πιο γρήγορα χάρη στο πρόγραμμα δράσεως των Βρυξελών σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες παρά τις σημαντικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των επιμέρους ΛΑΧ. Στην περίοδο 2001-2010, οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες ε, στην οικονομία του συνολικά παρουσιάζουν ανάπτυξη της τάξης του 6% κατά μέσο όρο κατέτος. Οι χώρες αυτές ε, παρουσιάζουν ανάπτυξη κυρίως προς το ΑΕΠ τους και προχωρούν ε, προς την ικανοποίηση των στόχων της, της χιλιετίας με την βελτίωση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στην πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό και κάποιους δείκτες ε, ισότητας των φύλων σε πολλές από τις χώρες που αποτελούν μια πολύ θετική ένδειξη από το 1990 για πρώτη φορά. Πολιτικές μεταρρυθμίσεις, εκδημοκρατισμός, διαφάνεια, βελτίωση του δικαστικού συστήματος στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες εν γέννη χαρακτηρίζονται από θετική εξέλιξη τα τελευταία δεκαετία. Οι ΛΑΧ παρουσιάζουν επίσης πρόοδο στην ε, χρηστή διακυβέρνηση, κυρίως όσον αφορά τις προσπάθειες για ε, εξασφάλιση και θέσπιση δημοκρατικών θεσμών και συμμετοχή στην εξουσία των γυναικών. Επίσης, οι αναπτυξιακοί εταίροι έχουν καταβάλει προσπάθειες να ε, προχωρήσουν στις ε, μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται από δική τους πλευράς. Έχουμε παραδείγμα βελτίωση στην ικανοποίηση του χρέους, χάρη και στην απαλλαγή από το χρέος που είχε χορηγηθεί με την ε, περίφημη πρωτοβουλία HIPIC και την πολυμερή απόφαση πρωτοβουλία για μείωση του χρέους, MDRI. Έχουμε σημαντική μείωση σε όγκο, 37 δολάρια ΗΠΑ για το 2008 δηλαδή, αν και το ποσοστό της διεθνούς χορηγίας ε, ήταν πολύ χαμηλό, ήταν κάτω από το 0,23% που είχε διεκδικήσει το πρόγραμμα δράσης των Βρυξελών. Στο εμπόριο, οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες μπόρεσαν να αξιοποιήσουν μια σειρά προτιμησιακών καθεστώτων και σχέσεων συναλλαγών, ε, παραδείγματι απαλλαγή από τελωνιακούς δεσμούς, από ποσοστώσεις, ε, πρόσβαση σε αγορές, σε αναπτυγμένες χώρες για τα προϊόντα τους. Πλην όμως είναι ακόμη πολύ δύσκολη η κατάσταση προς εξαγωγές λόγω των φραγμών στην είσοδο στην αγορά, μη τελωνιακών φραγμών δηλαδή, και επίπεδου, υψηλού επίπεδου των προδιαγραφών που απαιτούνται από τις ε, χώρες ε, προς οποίες θα μεταβούν αυτές οι εξαγωγές. Οι άμεσες επενδύσεις σε ροές βελτιώθηκαν από τα 6 δις δολάρια το 2000 στα 35 δις το 2008. Όμως οι περισσότερες επενδύσεις στοχεύουν την εξορυκτική, τον εξορυκτικό κλάδο και παρά τις θετικές εξελίξεις η αξιολόγηση ε, του προγράμματο δράση των Βρυξελών, στην οποία προβάλλουμε σήμερα, δείχνει ότι οι περισσότερε από τι λιγότερο ανεπτυγμένε χώρε δεν έχουν μπορέσει να φτάσουν στου στόχου που είχαν οριστεί με το πρόγραμμα δράση των Βρυξελών. Και ακόμη αντιμετωπίζουν σημαντικά ε, προβλήματα και προκλήσει ω προ την ανάπτυξη. Παραδοσιακέ προκλήσει, δηλαδή άκρα, φτώχεια, διαρθρωτικέ αδυναμίε, απουσία υποδομών και δυναμικού υποδομών, γεωγραφική μειονεκτικά, με μειονεκτική θέση, έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού κατάλληλου για ανάπτυξη του δυναμικού και αδυναμία αντιμετώπιση των εξωτερικών κλειδονισμών οδηγούν σε αδυναμία για τις χώρες αυτές να βελτιώσουν την ζωή των πολιτών τους. Οι νέες προκλήσεις και οι ευκαιρίες κύπτουν στο παγκόσμιο αναπτυξιακό πεδίο από το 2001 στη διάθεσή τους, όμως οι χώρες αυτές δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και ουσιαστικά να δρέψουν τους καρπούς που προσφέρουν αυτές οι νέες ευκαιρίες. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται σοβαρή, ρεαλιστική δράση και από πλευράς αυτών των ε, λιγότερων αναπτυχμένων χρόνων αλλά και των αναπτυξιακών τους εταίρων. Είναι μικρό το ποσοστό μείωσης του χρέους, χαμηλή δηλαδή η ρυθμή. Εξίσου, σημαντικό κίνδυνο αποτελούν οι δημογραφικές πιέσεις για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Αυτή τη στιγμή οι χώρες αυτές τις ομάδες, έχουν 880 εκατομμύρια πολίτες συνολικά. Με αύξηση όμως 2,3% θα έχουμε ε, πολύ υψηλό αριθμό νέων ανθρώπων στην αγορά εργασίας. Αυτό αποτελεί και πρόκληση αλλά και μεγάλη ευκαιρία οι λιγότερο ανεπτυγμένε χώρε θα χρειαστεί να εξασφαλίσουν τουλάχιστον 9,5, να εξασφαλίζουν τουλάχιστον 9,5 εκατομμύρια νέες θέσει εργασίας ανέτο, προκειμένου να διατηρήσουν την υφιστάμενη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασία, πράγμα που αποτελεί βέβαια τεράστιο εγχείρημα και παρότι ο γεωργικό τομέα είναι ο, ε, ο χώρο ο οποίο προσφέρει τι προστασίε εργασία στι χώρε αυτέ, η ικανότητά του για απορρόφηση εργατικού δυναμικού διαρκώ μειώνεται. Η γεωργική παραγωγικότητα παραμένει πολύ χαμηλή και αυτό επίσης το επιδεινώνει περαιτέρω η κλιματική αλλαγή ως φαινόμενο. Οι πρόσφατες και επάλληλες κρίσεις, στην, ε, οι επιστηστικές, στην ενέργεια, στα βασικά αγαθά, η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχουν βεβαίως αποδείξει πόσο ευάλωτες είναι αυτές οι χώρες στα εξωτερικούς κοινωνισμούς. Δεν μπόρεσαν δηλαδή να εξασφαλίσουν αυτό το μαξιλάρι ασφαλείας ε, που θα απορροφούσε τον κλειδονισμό τον εξωτερικό και επίσης απεδείχθη ότι οι φυστάμενοι ε, μηχανισμοί εξωτερικής βοήθειας που είχε προβλέψει το σχέδιο δράσης των Βρυξελών δεν ήταν επαρκείς για να στηρίξουν τις χώρες αυτές σε ένα επίπεδο ικανοποιητικό. Ξιότιμοι κυρίες και κύριοι, μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Αφού σας εξήγησα, σας έδωσα μια σύνοψη της αξιολόγησης του προγράμματος δράσης των Βρυξελών. Προχωρούμε τώρα προς την Ισταμπούλ με τον ίδιο περίπου αριθμό ε, λιγότερων αναπτυγμένων χωρών όπως το 2001. Δύο μόνο χώρες, το Πράσινο Ακροτήριο και οι Μαλδίβες, κατάφεραν να ξεπεράσουν ε, τα όρια της ομάδας αυτής μέσα στην δεκαετία που πέρασε. Είναι σημαντικό λοιπόν να ανανεωθεί η δέσμευση απέναντι στην συνεργασία με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και να υπάρξει νέο πρόγραμμα δράσης δημιουργία περαιτέρω συνεργασιών στον αγώνα κατά της στόχιας είναι σημαντικό για την τέταρτη διάσκεψη των Ηνωμένων Αθηνών για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Θα σας εξηγήσω ποια είναι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα. Οι προετοιμασίες για την τέταρτη διάσκεψη των λιγότερων αναπτυγμένων χωρών συνεχίζονται και μάλιστα με μια προσέγγιση από τα κάτω, ξεκινώντας από το επίπεδο της κάθε χώρας. Εθνικές διαβουλεύσεις διεξήχθησαν ολόκληρο το 2009 με συμμετοχή σημαντικού φάσματος ενδιαφερομένων μερών. Έγιναν και συναντήσεις περιφερειακής επανεξέτασης των θεμάτων στην Αφρική και στην Ασία με τη συμμετοχή των λιγότερων αναπτυγμένων χωρών και των αναπτυξιακών εταίρων τους στο παγκόσμιο επίπεδο το γραφείο μου, σε στενή συνεργασία με άλλες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και άλλους διεθνείς οργανισμούς, οργάνωσε έναν αριθμό εκδηλώσεων για διάφορα θέματα, σε διάφορες θεματικούς χώρους, με ιδιαίτερη σημασία για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. 13 από αυτές τις διοργανώσεις έχουν ήδη εξαχθεί και τρεις προγραμματίζονται για τις επόμενες ημέρες οι συνόψεις και τα απορίσματα των εκδηλώσεων αυτών θα χρησιμοποιηθούν ως εισρωές για τη δημιουργία του νέου προγράμματος δράσης. Πέραν τώρα από τη συνεργασία αυτή στο διακυβερνητικό επίπεδο, ακολουθούμε τρεις άλλες οδούς, κοινοβουλευτική, κοινωνία των πολιτών και ιδιωτικού τομέα. Έχουμε εργαστεί ήδη για να θεσπίσουμε μια στέρεα θεσμική βάση για αυτή αυτές τις τρεις οδούς που να παραμείνουν ενεργές και μετά από την εφαρμογή του νέου προγράμματος δράσεως. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών διόρισε ε, μια ομάδα σημαντικών προσωπικότητων για να εξετάσουν τα κολλήματα που αντιμετωπίζουν οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες στην ε, οικονομική τους πρόοδο, να συστήσει νέα υποδείγματα διαρθρωτικών ε, μεταρρυθμίσεων και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση, να δημιουργήσει στενούς δεσμούς συνεργασίας των λιγότερων ε, ε, αναπτυγμένων χωρών. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες θα σφυριλατήσουν τις συνέργειες μέσα στην προπαρασκευαστική φάση της διασκέψεως. Στο παγκόσμιο επίπεδο, ο διακυβερνητικός διάλογος και διαβούλευση έχουν ήδη αρχίσει. Η πρώτη συνάντηση της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής διεξήχθη τον Ιανουάριο στη Νέα Υόρκη Εκεί συζητήθηκαν τα στοιχεία ενός σχεδίου εγγράφου. Η δεύτερη συνάντηση της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής θα διεξαχθεί τον Απρίλιο και θα αποτελέσει το επόμενο στάδιο της σύνταξης του εγγράφου. Ορισμένες από τις προτεραιότητες που έχουν ήδη προταθεί στο τρέχον έγγραφο του νέου προγράμματος δράσεως περιλαμβάνουν και τις σημαντικές προκλήσεις τις οποίες εξήγησα προηγουμένως. Οι βασικές προτεραιότητες έχουν ως εξής. Πρώτο, δημιουργία ικανότητας παραγωγής στον αγροτικό, βιομηχανικό και τομέα υπηρεσιών και υποδομές. Δεύτερο, προώθηση της ανάπτυξης στον γεωργικό τομέα, τομέα ασφάλειας τροφίμων και αγροτικό. Τρίτο, προώθηση του εμπορίου με πρόσβαση στις αγορές, με αύξηση της δυνατότητας από πλευράς προσφοράς και ε, σταθεροποίηση τιμών. Τέταρτο, ενίσχυση της ανάπτυξης του ανθρώπινου και κοινωνικού δυναμικού, ισότητα των φύλων και ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών. Πέμπτο, αύξηση της ανθεκτικότητας απέναντι σε πολλαπλές κρίσεις και άλλες αναφιόμενες προκλήσεις. Έκτο, κινητοποίηση οικονομικών πόρων για την ανάπτυξη και για τη δημιουργία ικανοτήτων. Έβδομο, προώθηση της, της χρηστής διοίκησης και διαχείρισης στο εθνικό και διεθνές επίπεδο και στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αξιότιμοι ευρωβουλευτές, καθώς προχωρούμε σε μια νέα δεκαετία και σε μια νέα εποχή όπου είναι σαφής πλέον η αναγνώριση ότι οι 48 λιγότερα αναπτυγμένες χώρες έχουν ωστόσο και μεγάλο απόθεμα φυσικών πόρων και μπορούν να αποτελέσουν κινητήρια δύναμη και για την παραγωγική και για την κατανάλωση για να υλοποιηθούν οι υποσχέσεις παγκοσμιοποίησης, αλλά για να συμβεί αυτό χρειάζεται καταβολή ειδικών προσπαθειών στο διεθνές επίπεδο. Επιτρέψτε μου να έλθω τώρα στον ρόλο των βουλευτών στην υποστήριξη των λιγότερων ανεπτυγμένων χωρών για την εφαρμογή του νέου προγράμματος δράσεως και του προγράμματος δράσεως των Βρυξελών. Από την τρίτη διάσκεψη για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, η Διακοινοβουλευτική Ένωση και το δικό μου γραφείο έχουμε <clears throat> θεσπίσει μια καρποφόρο συνεργασία για την πρόθεση εφαρμογής του προγράμματος δράσεως των Βρυξελών στη δεκαετία 2009-2010. Ως ανέφερα προηγουμένως, οι βουλευτές των λιγότερων ανεπτυγμένων χωρών έχουν εμπλακεί στενά στην προπαρασκευαστική διαδικασία της τέταρτη διασκέψεως των Ηνωμένων Εθνών για τι λιγότερο αναπτυγμένε χώρε και στο εθνικό και στο περιφερειακό επίπεδο έχοντα <clears throat> συνεισφέρει για τον καθορισμό προτεραιοτήτων για την επόμενη δεκαετία αναπτύξεως. Οι δραστηριότητες <clears throat> της κοινοβουλευτικής διαστάσεως θα κορυφωθούν με την συνεργασία σε ένα κοινοβουλευτικό φόρουμ λίγο πριν από την τέταρτη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στις 8 Μαΐου 2011 στην Ισταμπούλ. Το φόρουμ αυτό θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ε, κοινοβουλευτικής διάστασης και του ενεργού ρόλου που θα παίξει στην συνέχεια και στην εφαρμογή του νέου προγράμματος δάσος. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε εκεί να εγκρίνουμε μια διακήρυξη η οποία θα αποτελέσει την βάση για το προσεχές νέο πρόγραμμα δράσεως. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στον ρόλο που μπορούν να παίξουν τα κοινοβούλια για την, για την υλοποίηση των ε, διεθνών ε, υποχρεώσεων και θα συμμετάσχει προσωπικά στο Κοινοβουλευτικό Φόρουμ της Ισταμπούλ. Μετά από την διάσκεψη αυτή, ελπίζω ειλικρινώς ότι οι βουλευτές θα συμμετάσχουν και στην εφαρμογή και στο follow-up του νέου προγράμματος δράσεως το... οι διεθνείς οργανισμοί θα συμμετάσχουν για να αυξηθεί η ικανότητα των κοινοβουλίων των λιγότερων επιμένων χωρών να συμμετάσχουν στην υλοποίηση του νέου προγράμματος δράσεως, το οποίο θα ενισχύσει τις ικανότητες να μπει το νέο πρόγραμμα δράσεως σε όλα τα εθνικά προγράμματα για να αυξηθεί ο εποπτικός του ρόλος επί των εκτελεστικών εξουσιών. Να δοθούν και τα απαραίτητα δημοσιονομικά κονδύλια για την υλοποίηση του νέου προγράμματος δράσεως. Αγαπητοί αξιότιμοι ευρωβουλευτές, εν προκειμένου επιτρέψτε μου να αναγνωρίσω την σημαντική συμβολή της Ευρώπης προς ε, τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Θα ήθελα πρώτα να αποτίσω φόρο τιμής στις ευρωπαϊκές αξίες και στο ενδιαφέρον που δείχνεται για τις φτωχότερες και πιο ευάλωτες χώρες για την διατήρηση της αξιοπρέπειας και για την διασφάλιση καλύτερης, καλύτερου μέλλοντος. Έχετε δείξει δείγματα γενοδορίας προς τις ε, λιγότερο αμπτυμένες χώρες έχετε φιλοξενήσει τις τρεις προηγούμενες διασκέψεις και έχετε λάβει ιδιαίτερα μέτρα όπως για παράδειγμα το Everything But Arms, η πρωτοβουλία οτιδήποτε εκτός όπλων. Έχετε άλλωστε αποδειχθεί ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των λιγότερων ανεπτυγμένων χωρών. Υπό το πνεύμα αυτό σας απευθύνω έκκληση να συνεχίσετε την προσπάθεια ευαισθητοποίησης των κοινοβουλίων σας για τα σημαντικά αυτά θέματα. Δεύτερον, να κινητοποιήσετε την κοινή, τις κοινέ γνώμες ε, ε, πριν από την τέταρτη διάσκεψη που θα γίνει τέλη Μαΐου στην Ισταμπούλ. Τρίτο, να κινητοποιήσετε κονδύλια και υποστήριξη για την υλοποίηση του νέου προγράμματος δράσεως, περιλαμβάνοντας τις προτεραιότητες των λιγότερων ανεπτυγμένων χωρών σε όλες τις ε, κατανομές κονδυλίων. Και τέταρτο, να υποστηρίξετε την αύξηση των ικανοτήτων των κοινοβουλίων των λιγότερων ανεπτυγμένων χωρών για να υλοποιήσουν στο εθνικό τους επίπεδο πλέον το νέο πρόγραμμα δράσεως. Θα ήθελα τέλος να σας παρακαλέσω τι ευρωπαϊκές χώρες να μην αφήσετε τις παρούσες δυσκολίες που αντιμετωπίζετε να θαμπόσουν το όραμά σας για το μέλλον σχετικά με τη συνεργασία με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Συνεχίστε τη συνεργασία με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες γιατί αυτή θα αποβεί και προς όφελος της Ευρώπης συμβάλλοντας στην υπέρβαση της κρίσης. Υπολογίζω στην υποστήριξή σας για να αποβεί επιτυχία η τέταρτη διάσκεψη για τις λιγότερο ανεκτημένες χώρες. Ελπίζω επίσης ότι θα μπορέσετε να ενισχύσετε και να λάβετε μέτρα υποστήριξης της επόμενης δεκαετίας που θα ξεκινήσει με την διάσκεψη που θα γίνει στην Ιστανμπούλ για να εκπληρωθούν τα οράματα για τη μελλοντική ανάπτυξη των λιγότερων αναπτυγμένων χωρών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Merci, Σας ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε εδώ μαζί μας και επειδή μας κάνατε αυτό τον απολογισμό του προγράμματος δράσης σας, θα ήθελα να σας πω ε, τι διδάγματα έχετε αντλήσει από το πρόγραμμα δράσης. Ποιες είναι οι προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας και του προγράμματος που θα συσταθεί στην Κωνσταντινούπολη. Πώς αποτιμούμε το πρόγραμμα του παρελθόντος. Επίσης, ε, μιλήσατε και την αύξηση της εξωτερικής άμεσης επένδυσης αλλά περισσότερο αφορά τις εξορρυκτικές βιομηχανίες. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο αυτό έχει δημιουργήσει μία τοπική μορφή ανάπτυξης ή κατά πόσο ε, είχε επιπτώσεις στις χώρες αυτές. Ο κύριος Μπέρμαν. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω ευχαριστήσω τον ομιλητή για αυτή την συνεκτική παρουσίαση. Να ευχαριστήσω τον κύριο Σίτι γιατί ε, μιλήσατε για πολλούς τομείς παράλληλα. Μιλάτε για μια εκστρατεία ενσυνειδητότητα στις χώρες μας, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο όπως καταλαβαίνετε, διότι υπάρχει μεγάλη λιτότητα από πλευράς προϋπολογισμού, όπως είπατε και εσείς, και θα πρέπει να λογοδοτούμε για την δαπάνη των ε, χρημάτων και πολλά δεν βαίνουν καλώς και σε αυτόν τον τομέα. Δεν επιτυγχάνουμε τα αποτελέσματα που θα θέλαμε πάντα. Οι αναπτυξιακές πολιτικές βρίσκουν μια μεγάλη τροχοπέδη σε, ως προς θέματα γεωστρατηγικής σκοπιμότητας. Γνωρίζουμε ότι πολλοί δικτάτορες της Αφρικής είχαν παραμείνει στην εξουσία για αρκετές δεκαετίες και δεν τους ενδιέφερε η αναπτυξιακή πολιτική αλλά τα γεωστρατηγικά πολιτικά συμφέροντα και η ανάπτυξη φιλετικών καθαρά συμφερόντων. Άρα η αναπτυξιακή βοήθεια δεν ήταν επικοδομητική πάντα. Χρειάζεται, νομίζετε, μία ειδική στρατηγική και προσέγγιση σε σχέση με τα ευάλωτα αυτά κράτη, όπου επικεντρώνεται η φτώχεια και η βία. Ίσως θα πρέπει να εστιάσουμε την αναπτυξιακή βοήθεια στις ΛΑΧ, προς τις ΛΑΧ θα πρέπει να εστιάσουμε προς τα εκεί την προσοχή μας και πιστεύετε ότι οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες θα ήταν η καλύτερη επιλογή. Η UNICEF τίνει να απαντήσει καταφατικά, διότι τα αριθμητικά στοιχεία θεωρούν ότι κάθε ευρώ ή κάθε δολάριο που επενδύεται είναι πιο αποτελεσματικό στην ανακούφιση της φτώχειας σε σχέση με χώρες που έχουν λίγο υψηλότερα εισοδήματα. Τώρα, ως προς τα γεωστρατηγικά συμφέροντα, πιστεύετε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου ε, λειτουργήσαν πραγματικά. Εγώ νομίζω ότι τα αποτελέσματα ήταν πενιχρά. Δεν θεωρείτε ότι αυτή η κοινωνική βόμβα στη Βόρεια Αφρική που εκρήγνει και τώρα μας δείχνουν ότι ήταν μεγάλο λάθος το ότι είχαμε αγνοήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Έχω ε, πολλές άλλες ερωτήσεις, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να παραμείνω εδώ. Ο κύριος Μίτσελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, θα ήθελα και εγώ να ε, καλωσορίσω τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Εγώ ε, βρέθηκα στην ενδιάμεση αναθεώρηση των Ηνωμένων Εθνών ε, επί του θέματος Εκ των υστέρων είδα ότι υπήρχε ένα ζωηρό ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση των ΛΑΧ και να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στους στόχους το, ως προς τις ΛΑΧ. Αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες στην Ευρώπη, διότι στη χώρα μου τον 19ο αιώνα αντιμετωπίσαμε τον λοιμό και το θέμα της ανάπτυξης έχει μεγάλη σημασία σε εμάς. Πολλές φορές στην Ιρλανδία συζήτησα και για παρηγορητική βοήθεια αλλά και για καθαρά αναπτυξιακή. Το είχα συζητήσει πρόσφατα με μία ε, συμπολίτη μου. Εάν λέμε στους ανθρώπους τα κακά νέα και το τι αρνητική επίπτωση έχουν, τότε θα καταβληθούν κάπως. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε μέρα πεθαίνουν 22.000 παιδιά, αλλά ε, και αυτό το ποσοστό κατέβηκε από τις 36.000 που είχαμε παλαιότερα. Άρα θα πρέπει να μιλάμε για ιστορίες επιτυχίας και όχι αποτυχίας. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε αυτό όταν επικεντρωθούμε σε κάτι. Μιλάμε γενικά για θέματα ισότητας ε, μεταξύ ανδρών και γυναικών. Μιλάμε για διατροφική ασφάλεια, θεματικά προγράμματα, γεωγραφικά προγράμματα. Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα στην έκθεσή μου. Ο κύριος Ντίβα έχει ε, διανύμει μια επιστολή του αναπληρωτή Υπουργού Άντρου Μίτσελ της Μεγάλης Βρετανίας όπου μιλάμε για, ε, για παιδιά που θα μπορούν να παρακολουθήσουν το σχολείο, μιλάμε για 11 εκατομμύρια, μιλάμε για ένα πρόγραμμα εμβολιασμού υγείας, να σώσουμε 50.000 γυναίκες που ε, γνωρίζουν επισφαλή ε, εγκυμοσύνη, να βοηθήσουμε της οικογένειας μέσα στα πλαίσια ενός οικογενειακού προγραμματισμού και ούτω καθεξής. Εάν δεν έχουμε ειδικού στόχους, κανείς τότε δεν λογοδοτεί. Πολλές φορές θεωρώ σε αυτή την ε, επιτροπή και σε άλλες επιτροπές θεωρώ ότι δεν κάνουμε τίποτα όταν μιλάμε με γενικόλογα. Δηλαδή, σε 10 χρόνια θα λέμε ότι πεθαίνουν 22.000 παιδιά που πεθαίνουν κάθε μέρα ή θα πρέπει να κατεβάσουμε το επίπεδο στους ε, στόχους στην θνησιμότητα της Ευρώπης. Νομίζω ότι και εσείς ε, θα πρέπει να μιλάτε για συγκεκριμένους στόχους, διαφορετικά δεν ε, επιτυγχάνουμε τίποτα και κανείς δεν λογοδοτεί, ούτε τα Ηνωμένα Έθνη ούτε κανείς άλλος. Ο κύριος Κόρτες Λάστρα. Κύριε Ντιάρα, χαίρομαι που είστε εδώ. Η παρουσία σας είναι πολύ σημαντική για την Επιτροπή μας, έτσι ώστε να δούμε τι στοιχεία έχουμε μέσα στα πλαίσια αυτής της τέταρτης διάσκεψης. Ελπίζουμε σε πολλά αποτελέσματα, είμαστε ρεαλιστές, αλλά θέλουμε αποτελέσματα για το μέλλον. Βεβαίως η ΛΑΧ πλήττονται περισσότερο από την μεγάλη αυτή κρίση και μέσα στα πλαίσια της διατροφικής ασφάλειας. Γι' αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί τουλάχιστον εν μέρη αυτό το πρόβλημα. Βεβαίως, η, ο περιορισμός της κρίσης σημαίνει ότι οι προϋπολογισμοί μας διαθέτουν λιγότερα χρήματα προς ε, την αναπτυξιακή βοήθεια. Δηλαδή μιλάμε για αναπτυξιακή βοήθεια γενικά, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει συντονισμός με τον απότερο στόχο των εργασιών μας. Μιλάμε για μεγαλύτερη αναπτυξιακή ασφάλεια ανά τον κόσμο. Οπωσδήποτε χρειάζεστε τη βοήθειά μας, χρειαζόμαστε ένα συντονισμό. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στην τέταρτη διάσκεψη και θα ήθελα να ρωτήσω το ίδιο που είπε και η κυρία Κέλλερ. Δηλαδή, με βάση την πείρα σας, πώς έχει η διαχείριση του προγράμματος, δηλαδή ποιο είναι το σημείο κλειδί, πώς μπορούμε να φτάσουμε σε καλύτερα αποτελέσματα στα πλαίσια αυτής της τέταρτης διάσκεψης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκέρενς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Διάρα για την παρουσία του και να τον ευχαριστήσω διότι αναφέρθηκε στο κοινοβουλευτικό φόρουμ που θα λάβει η χώρα πριν από τη διάσκεψη. Θα πρέπει να συνέλθουν και τα μέλη αυτά του φόρουμ έτσι ώστε να βοηθήσουμε περισσότερο τις ΛΑΧ πριν από την διάσκεψη. ήσασταν ιδιαίτερα αισιόδοξο κατά την αρχική σας παρουσίαση ως προς την έκβαση αυτής της διάσκεψης, αλλά πέρα από τις κοινοτοπίες που αναφέρονται, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μία σειρά από αλήθειες. Δηλαδή, να μην ξεχνάμε ότι πρέπει να πούμε πολλές αλήθειες στις ΛΑΧ, αλλά και εκείνες πρέπει να μας πούν, να πούν προς εμάς πολλές αλήθειες. Θα πρέπει να προβούμε και σε μία αυτοκριτική, δηλαδή δεν ε, ανταποκριθήκαμε στις δεσμεύσεις μας της τάξης του 0,7%. Δηλαδή βρισκόμαστε έτη φωτός μακριά από τους αρχικούς στόχους. Αυτό είναι σκανδαλώδες, θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να επιτευχθεί συνένεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο με βάση τους αναπτυξιακούς στόχους που είχαν τεθεί το 2005. Θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς σε, ως προς αυτό το σημείο και να μιλήσουμε και για ένα συμπληρωματικό ε, κόστος το οποίο θα πρέπει να υπομισθούμε για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών ως προς τις δηλώσεις του, του Παρισιού θα πρέπει να συμβαδίζουμε με τους στόχους μας. Sur les relations et les pays émergents. Euh, και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο υπάρχει αμφισημία ως προς τους στόχους με βάση τις ε, δηλώσεις του Παρισιού και της δακάρ, Διότι υπάρχουν ε, οι αναδιόμενες χώρες οι οποίες βεβαίως δεν συγκαταλέγονται ούτε, στο, ούτε στις ΛΑΧ αλλά ούτε και στις χώρες μέσου εισοδήματος. Δηλαδή μέσα στα πλαίσια του ΠΟΕ θα πρέπει να προβούμε σε μία βοήθεια προς τις ε, λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Οι αναδυόμενες χώρες όμως ήταν αυτές που οδήγησαν στην αποτυχία των συμφωνιών μέσα στα πλαίσια ας πούμε των εισαγωγών ε, μπανάνας από τις ΛΑΧ. Δηλαδή οι αναδυόμενες χώρες με το σιγοντάρισμα των Ηνωμένων Εθνών ήταν αυτές που έθεσαν τέλος στα πλεονεκτήματα τα οποία γνώριζαν οι χώρες ΑΚΕ. Αυτές τις ε, αμφισημίες θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Όσοι βρεθήκατε στο Χόνγκ Kong τις διαπραγματεύσεις για την αναδιάρθρωση του παγκοσμίου εμπορίου, είδατε ότι οι Αφρικανοί στην ουσία πολτοποιήθηκαν από τις αναδυόμενες χώρες θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και αυτό το σκέλος του θέματος. Επίσης θα πρέπει να μιλήσουμε για τις θεσμικές ασυμμετρίες. Ένας ε, από τους λόγους για τους οποίους σας υποστηρίζουμε είναι επειδή αντιμετωπίζεται μία ε, θεσμική αδυναμία εναντί του ΠΟΕ. διότι όταν εγκριθούν αυτά τα μέτρα από τα κράτη-μέλη, τα μέτρα αυτά είναι δεσμευτικά Διαφορετικά, κανείς μπορεί να προσαχθεί ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου Επίλυσης Διαφορών. Οι δικές σας αποφάσεις δεν είναι δεσμευτικού χαρακτήρα. Είναι καθαρά ακαδημαϊκού ή συμβουλευτικού. Εάν θέλουμε να βοηθήσουμε τις λιγότερο αναπτυγμένε χώρες, θα πρέπει αυτές οι συστάσεις να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, δηλαδή του Διεθνούς Γραφείου εργασία. Μέσα στα πλαίσια της νέας διακυβέρνησης που δημιουργείται, θα πρέπει να δώσουμε τέλος την ε, απουσία των ΛΑΧ σε όλα τα διεθνή φόρα. Στα πλαίσια των ε, G20 δεν το είδαμε αυτό το κεφάλαιο. Μιλάμε για ένα 80% του παγκόσμιου ΑΕΠ που ε, εκπροσωπούν οι χώρες των, των G20, αλλά το υπόλοιπο 20% δεν εκπροσωπείται καθόλου και ιδιαίτερα η ΛΑΧ. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ επιθετικοί στην προσέγγιση μας σε σχέση με, τα, ε, με τη διάσκεψη αυτή της Κωνσταντινούπολης βεβαίως. Πολλές φορές ε, είναι κανείς επιφυλακτικός. Αν θέλετε όμως να προβάλλουμε μία ε, στεναρή θέση, να προβάλλετε μάλλον, μπορούμε να σας βοηθήσουμε και εμείς μέσα στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού φόρουμ ιδιαίτερα. Έτσι ώστε το μήνυμα αυτό να περάσει προς τους ενδιαφερόμενους υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι. Σας υποστηρίζουμε στεναρά μέσα στα πλαίσια των πολυμερών σχέσεων και θα πρέπει να συνεισφέρουμε στην ε, σοβαρή, στη σοβαρή σας εργασία. Και τέλος, το πράσινο ακροτήριο δεν ε, εντάσσεται πλέον στις ΛΑΧ Το πράσινο ακροτήριο βγήκε λοιπόν από την κατηγορία του ΛΑΧ και δεν γνωρίζει, δεν ε, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το προτιμησιακό καθεστώς που μπορούσε να έχει το πράσινο ακροτήριο όταν εντασσόταν στις χώρες ΛΑΧ. Δηλαδή ε, αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι για ορισμένες χώρες γιατί μερικές φορές υπάρχει μερική πρόοδος, αλλά όχι επαρκής. Ο κύριος Ντέβα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ το Γενικό Γραμματέα. Ήταν πληρέστατη η παρουσίαση των στόχων. Θα αναφερθώ σε τρία διαφορετικά θέματα. Καταρχάς, θεσμικά, και εδώ θα ήθελα να επισημάνω την προσοχή σε ορισμένα ζητήματα. Ο κ. Μίτσελ, ο φίλος αναφέρθηκε στο γεγονό ότι υπάρχουν κάποιε επιφυλάξει, ε, Δεν θέλουμε να πηγαίνουμε στην ε, διάσκεψη. Εγώ αρνήθηκα προσωπικώ να πάω στη Νέα Υόρκη. Γιατί? Σε προηγούμενε εκδηλώσει, ο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου στη Νέα Υόρκη ήταν ε, αποτροπιαστικό. Εμεί είμαστε ισότιμα μέλη εδώ μέσα από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε κάποια δομή υπουργική, δεν ακολουθούμε τις δομές των κρατών μελών. Είμαστε ίσοι με την Επιτροπή και το Συμβούλιο, δυνάμει της συνθήκης της Λισαβόνας. Έχουμε συνομοθετικές αρμοδιότητες. Η Επιτροπή είναι ένα εκτελεστικό όργανο. Εμεί είμαστε η αρχή αρμόδια για τον προπολογισμό. Εμεί δεν θέτουμε τα χρήματα. Έχουμε την ευθύνη για τον προπολογισμό και με οφείλουμε και να εξηγούμε στο φορολογούμενο τι τα κάναμε τα χρήματα που διαθέσαμε. Και μια πολύ σημαντική και υπάρχει μια πολύ σημαντική δομή, η δομή δηλαδή με την οποία η Επιτροπή μας εξηγεί τι έκανε με τα χρήματα αυτά. Άρα, εάν μπορώ να το πω έτσι κομψά, γίνεστε με, μέσω αυτή τη δομή. είστε κάποιοι από τους υπηρέτες μας, κάνετε αυτό που έχουμε δώσει εμεί εντολή να γίνει. Αλλά και εγώ βέβαια πρέπει να εξηγήσω μετά στο φορολογούμενο το τι έχω κάνει με τα λεφτά του. Άρα λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό το να δίδεται λογαριασμό, το να υπάρχουν στόχοι, το να, υπάρχουν, το να επιτυγχάνονται οι στόχοι και το να συμμετέχουμε και εμείς στο ύψιστο δυνατό επίπεδο για να συνεχίσει να ρέει το χρήμα. Διότι αν δεν συμμετέχουμε εμείς σε αυτές τις εκδηλώσεις και δεν μπορούμε να εξηγήσουμε στο προλογούμενο ότι έχει γίνει, Όπω λέγεται και στην έκθεση μου, υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία τώρα ο, ο φορολογούμενο δεν θέλει τη χρηματοδότηση, γιατί πια έχει κόποση χρηματοδοτική. Αυτό είναι το θεσμικό θέμα, μας το στο οποίο θέλω να αναφερθώ. Το δεύτερο, πριν από 10 χρόνια με τον Μασκάλα Μη και κάποιους άλλους που ακόμα είναι εδώ παρόντες, ξεκινήσαμε την πρωτοβουλία «Τα πάντα πλην όπλων» για, τις, ε, για την ενίσχυση από ευρωπαϊκής ε, πλευράς προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Τελικά έγινε anything but farms, τα πάντα πλην των γεωρικών προϊόντων. Δηλαδή του επιτρέπαμε να, εισάγουν, να εξάγουν μάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι γεωργικά προϊόντα. Και με χαρά άκουσα σήμερα από εσά ότι θα συζητηθούν με το βάση το πρόγραμμα της διάσκεψης και τα γεωργικά ε, προϊόντα. Γιατί βέβαια οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες τι έχουν να προσφέρουν. Δεν έχουν ούτε κομπιούτερ, ούτε υψηλή τεχνολογία, ούτε παραγωγή λογισμικού, ούτε βαριά βιομηχανία, γεωργικά προϊόντα έχουν να προσφέρουν. Ερωτώ λοιπόν, με την πρωτοβουλία τα πάντα πλην όπλων, τι έχουμε καταφέρει, ή εν πάση τα πάντα πλην γεωργικών. Θέλω στοιχεία, στόχους, επιτεύγματα. Υπάρχει κάτι τέτοιο να μας δώσετε. Και τρίτον, δυστυχώς, η ΛΕΑΧ έχουν να αντιμετωπίσουν το στόχο της ενίσχυσης της οικονομικής τους, δηλαδή τη δημιουργία πλούτου. Ταυτόχρονα όμως έχουν και τις χειρότερες δομές όσον αφορά και τη δημιουργία, ε, η σύσταση εταιριών, την ε, ε, κατάρτιση καταστατικών, εγγραφή, θέσπιση. Όταν χρειάζονται 20 μήνες για να θεσπιστεί μια εταιρεία με όλη τη γραφειοκρατία που επικρατεί εκεί, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να παραγάγουν πλούτο. κυρία Ζωλή. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Θεοχάρου τελευταία. Ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε. Your Excellency, I'm going to speak in Greek, so please use your headphones. Uh, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Διάρα για την ενδιαφέρουσα ομιλία σας. Συγχωρέστε μου την άγνοια, αλλά ήθελα να ρωτήσω τρία συγκεκριμένα πράγματα. Αυτές οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες έχουν εμπλακεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας σε πολέμους, είτε μεταξύ τους είτε με άλλες χώρες. Έχουν εμπλακεί σε εξοπλιστικά προγράμματα και διαθέτουν μεγάλα κονδύλια από το εισόδημα τους για την αγορά όπλων. Και ένα τρίτο ερώτημα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία αν η διαφυγή επιστημόνων και εξειδικευμένων επαγγελματιών από αυτές τις χώρες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε, μειώθηκε, συνεχίζεται, είναι σταθερή. Όλα αυτά τα ζητήματα θα συζητηθούν στην Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης. Υπάρχουν συγκεκριμένα κεφάλαια στα οποία θα μπορούσε κάποιος να στηρίξει θέσεις συγκεκριμένες επί των ζητημάτων τούτων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Craig McCann από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για πέντε μόνο λεπτά, γιατί έχουμε καθυστερήσει πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Με χαρά λαμβάνω το λόγο στο θέμα αυτό. Ονομάζομαι Peter Craig McQuaid, όπως είπατε και εσείς, είμαι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ για τη σχέση με, τα Ηνωμένα Έθνη και την προετοιμασία της διάσκεψης, της τέταρτης διάσκεψης. Με χαρά βλέπω και τον κύριο Σέκτη Σιντιντιάρα σήμερα για την προετοιμασία της διάσκεψης και την κατάσταση των ΛΑΧ. Θα συμφωνήσω με πολλά από τα σχόλια που ακούστηκαν και από τον κύριο Σιτιτιάρα και από τους παρευρισκόμενους βουλευτές. Επιτρέψτε όμως να σας δώσω κάποιες πληροφορίες για τις δικές μας ε, προετοιμασίες για ε, τη συμμετοχή σε αυτή τη διάσκεψη εκ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ένα έγγραφο βάσης ε, που έχει προετοιμάσει η Γενική Γραμματεία και βέβαια έχουμε να παρουσιάσουμε και τις θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης στην συνεργασία με το Συμβούλιο. Ήδη σήμερα σε επίπεδο ομάδας εργασίας για την ανάπτυξη συζητείται ακριβώς η τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέταρτη διάσκεψη. Έχουμε θεσπίσει και το έγγραφο εργασίας 16 Φεβρουαρίου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις θέσεις Επιτροπής και το, το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών πιστεύουμε πολύ στόμα θα εγκρίνει τη σχετική θέση Ευρωπαϊκής Ενώσης πάλι εν ώψη της ίδιας της διάσκεψης. Για να περιγράψω με αδρές γραμμές ε, τις θέσεις μας, υποστηρίζουμε βεβαίως τους στόχους ε, της ε, αναγωγής ε, ε, των χωρών αυτών λάχα ώστε να βγουν από την κατηγορία λάχ μέχρι το τέλος της δεκαετίας χρειάζονται πιο, πιο συστηματικοί μηχανισμοί και συγκεκριμένες χρονικές ε, χρονικά κριτήρια ώστε να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να ανέβουν επίπεδο, να ξεφύγουν δηλαδή από το επίπεδο των λάχα κάνουμε κι εμεί από πλευρά μα ό,τι μπορούμε για να τα στηρίξουμε με τι διάφορε πτυχέ στήριξη, είτε σε ενίσχυση είτε, εμπορικά, είτε με εμπορικά μέτρα. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει και οι χορηγοί να συνεχίσουν να προσπαθούν για τους στόχους 0,85 85-0,2 ε, για την βοήθεια προς τις ε, λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Πρόκειται για μια δέσμευση την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επαναλάβει από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε ότι η ανάπτυξη είναι κοινή πρόκληση, αλλά στο με δεδομένη αυτή την πρόκληση κύρια ευθύνη για την ανάπτυξη των ΛΑΧ έχουν οι δικέ του κυβερνήσει, αυτέ οι κυβερνήσει δηλαδή οι ίδιε. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να κοιτάξουμε από την εμπειρία που έχουμε ε, στην επίτευξη αυτών των αναπτυξιακών στόχων από κάποιε χώρε, ποιε είναι εκείνε που είναι πιο επιτυχεί, που υπάρχουν κάποιε, υπάρχουν και αρκετά στοιχεία, ε, κείμενα, μελέτε και από, τις Ηνωμένα, από τα Ηνωμένα Έθνη για τι χώρε που μπόρεσαν και οικονομική ανάπτυξη αλλά και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού να εξασφαλίσουν με καλέ πολιτικέ και όχι μόνο μόνο με την βοήθεια την εξωτερική, δηλαδή την βοήθεια ή τη χορηγία από άλλους παράγοντες. Πιστεύουμε ότι πρέπει να βελτιωθούν, να ενισχυθούν και να βελτιωθούν οι φυστάμενοι μηχανισμοί και να ενισχυθούν και οι φυστάμενε δεσμεύσει για τις ΛΑΧ. Κάθε πηγή χρηματοδότηση θα πρέπει να αξιοποιηθεί και όχι μόνο η βοήθεια. Οι αναδυόμενες οικονομίες και δεδομένου του μεταλλασσόμενου οικονομικού σκηνικού έχουν και αυτές καθήκον να προσφέρουν στήριξη σε αυτές τις ε, χώρες, τις λιγότερο ανεπτυγμένες. Η στόχευσή μας θα πρέπει να πηγαίνει περισσότερο προς το αποτέλεσμα και με βάση και την τελευταία διάσκεψη του Σεπτεμβρίου πιστεύουμε ότι υπάρχουν τρία ζητήματα που θα πρέπει να στηθούν, το πόσο ευάλωτε και τα στρωτά σημεία αυτών των χωρών και οικονομικά αλλά και άλλα όπως φερειπίν συγκρούσεις. Δεύτερον θα πρέπει να οικοδομηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την βιώσιμη ανάπτυξη των ΛΑΧ και τρίτον με δημιουργία αυτού του περιβάλλοντος θα πρέπει να προωθήσουμε την ανάπτυξη στις ΛΑΧ με, μια, ε, με τρόπο συνεκτικό και συμπεριληπτικό ε, με αυτές λοιπόν τις τρεις, ε, αυτά τρία κριτήρια έχουμε ετοιμάσει προτάσεις για τα κράτη-μέλη που πιστεύουμε θα ε, είναι ικανοποιητικές, θα γίνουν δεκτές και με βάση αυτές θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και ίσως και με προτάσεις από πλευρά των κρατών μερών θα προχωρήσουμε προς την διάσκεψη. Αφού ολοκληρωθούν βέβαια οι διαδικασίες του Συμβουλίου σε κανένα δύο εβδομάδες. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα το λόγο θα λάβει ο κύριος Σιντιντιάρα για να απαντήσει για οκτώ λεπτά παρακαλώ. Like Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σχολιάσω καταρχήν τα όσα είπε η κυρία Κέλλερ. Ποια είναι τα διδάγματα που αντλήσαμε, τι λειτουργεί και τι όχι. Αν και έχει επιτελεστεί πρόοδος, όπως σας είπα, με βάση τις αρχικές δεσμεύσεις των εταίρων, για τη μείωση του χρέους, πρόσβαση στις αγορές, άμεσες επενδύσεις, αύξηση των εμβασμάτων που προέρχονται από τους μετανάστες, καλύτερη διακυβέρνηση καλύτερη κινητοποίηση, χρήση των εγχώριων πόρων, μιλάμε για ένα 23% του ΑΕΠ, παρόλα αυτά υπάρχουν μεγάλες αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, η φέρπη, η φτώχεια και η οικονομική ανάπτυξη της τάξης του 6% δεν αντικατοπτρίζεται στο μέσο πολίτη οι επενδύσεις, ιδιαίτερα στην εξορυκτική βιομηχανία, δεν έχουν έναν διαφορετικό δεσμό με την υπόλοιπη οικονομία. Υπάρχει δηλαδή συμμετοχή μιας ελίτ και μόνο. Όλα αυτά θα πρέπει να αλλάξουν. Θα πρέπει να έχουμε μία βιώσιμη ανάπτυξη και συμπεριληπτική, αν θα μπορούσα να πω. Έτσι ώστε το κράτος να έχει τη δυνατότητα παρέμβασης πέρα από το ρυθμιστικό του ρόλο, έτσι ώστε να επικρατήσει η ισότητα ως προς τον επιμερισμό του πλούτου, της δημιουργίας ευκαιριών για τους πολίτες και ούτω καθεξής γιατί ο ιδιωτικός τομέας και επενδύσεις από μόνες τους δεν μπορούν να δημιουργήσουν ισότητα και δικαιοσύνη. Χρειάζεται κρατικός παρεμβατισμός. Από ό,τι μάθαμε από τις Βρυξέλλες είναι ότι πρόκειται για έναν εκτενή μηχανισμό. Γιατί η αναπτυξιακοί στόχοι της ε, χιλιετίας δεν είναι παραδείκτες πώς να καταπολεμήσουμε το λοιμό, τις ασθένειες, να παρέχουμε σχολεία για τα παιδιά, αλλά η αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας δεν ε, οδηγούν προς μία κινητοποίηση γιατί από τις Βρυξέλλες μάθαμε πώς ε, κινούνται αυτοί οι μηχανισμοί, πώς λειτουργούν αυτοί οι μηχανισμοί. Το πρόγραμμα των Βρυξελών όμως ήταν πολύ φιλόδοξο. Ε, θέλησε να καταπολεμήσει κάθε είδος ευαλωτότητας. Επίσης δεν υπήρχε ένας μηχανισμός, ένας ελεγκτικός ή εποπτικός μηχανισμός που να ελέγχει τις ΛΑΧ και τους εταίρους. Άρα, πρόθεσή μας είναι να εστιάσουμε την προσοχή μας σε συγκεκριμένες θεματικές στην Κωνσταντινούπολη. Και εγώ θα προτιμούσα το εξής. Ό,τι και να μας απασχολήσει στους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας θα πρέπει να έχει καθαρά εποπτικό ρόλο και να εστιάσουμε την προσοχή μας σε επιμέρους θέματα που αφορούν τις ΛΑΧ. Δηλαδή την διαρθρωτική ευαλωτότητα τη... και... και την έλλειψη βασικών υποδομών όπως και παραγωγή ενέργειας. Θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε τρεις-τέσσερις τομείς για να δούμε τι μπορούμε να επιτύχουμε για την επόμενη δεκαετία. Και θα προσπαθήσω να πείσω τα κράτη-μέλη να το επιτύχουν αυτό. Ε, κύριε Μπέρμαν, συμφωνώ με το, με το θέμα της λογοδοσίας. αυτό είναι καλύτερος, ο καλύτερος τρόπος έτσι ώστε οι φορολογούμενοι στη, από τις χώρες δωρητές να ξέρουν πού πηγαίνουν τα χρήματά τους και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Γι' αυτό θα προβάλλουμε έναν ε, στεναρό, έναν δυνατό μηχανισμό που θα αφορά την σχέση δωρητών παραληπτών. Δηλαδή να έχουμε ένα μηχανισμό follow-up, ένα μηχανισμό παρακολούθησης ή για να ξέρουμε τι επιτελέστηκε, τι όχι και ποια ήταν η επίπτωση της βοήθειας στις ε, παρεμβατικές αυτές δράσεις. Ως προς τη χρήση πόρων από τους δικτάτορες της Βορείου Αφρικής. Αυτό το αφήνω σε εσά. Θα το κρίνετε εσείς. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως, ότι οι περισσότερες χώρες της Βορείου Αφρικής δεν είναι λάχ οι ΛΑΧ αφορούν την υποσαχάρια περιοχή, όπου υπάρχουν και θέματα διακυβέρνησης που θα πρέπει να μας απασχολήσουν για να υπάρχει διαφάνεια. Θα πρέπει να εστιάσουμε τη χρήση πόρων στις ΛΑΧ, γιατί είναι οι χώρες που υπολείπονται και βρίσκονται πολύ πίσω ως προς τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας. Άρα, η βιώσιμη ανάπτυξη θα πρέπει να είναι ε, ένα είδος λογοτύπου για τις ΛΑΧ. Άμεση εξωτερική επένδυση λοιπόν. Αυτή είναι η λέξη κλειδί, αλλά αυτό θα πρέπει να σημαίνει ότι δημιουργούμε κίνητρα και στις χώρες προέλευσης έτσι ώστε να δουν τις δυνατότητες, το δυναμικό αυτό των ΛΑΧ. Ο κύριος Μίτσελ μιλά για στοχοθέτηση. Βεβαίως, σας είπα ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι είναι πολύ συγκεκριμένοι ποσοστή αναλογία παιδιών που πάνε στο σχολείο, ισότητα των δύο φύλων, θέμα διατροφικής ασφάλειας, μείωση φτώχειας, μείωση θνησιμότητας των παιδιών και των ε, μητέρων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην ετήσια έκθεση των Ηνωμένων Εθνών Εκεί ακριβώς έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για το τι έχει επιτευχθεί μέσα σε ένα χρόνο. Αυτές οι πληροφορίες είναι πολύ σημαντικές. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο στη διάθεσή μου. Θα σταματήσω εδώ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε το λόγο σήμερα και βασιζόμαστε στην παρουσία σας στην Κωνσταντινούπολη Χαιρόμαστε διότι θα βοηθήσετε τις ΛΑΧ πέρα από τις εγγενείς δυσκολίες που γνωρίζετε και εσείς. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντιάρα. Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε στο θέμα 12 της ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για ένα από τα μεγάλα μέσα των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας και των μηχανισμών αναπτυξιακής συνεργασίας και θα δώσω το λόγο στον κύριο Μίτσελ για να μας μιλήσει για το, τον πολιτή χαρακτήρα αυτού του μέσου. Ευχαριστώ. Το DCI, ο Μηχανισμός Αναπτυξιακής Συνεργασίας, θα ισχύσει μέχρι το τέλος του 2013. Θα πρέπει όμως να κοιτάξουμε πέρα από αυτή την ημερομηνία. Η Κομισιόν θα υποβάλει προτάσεις για μετά το 2013 για το πολιετές οικονομικό πλαίσιο πριν από το καλοκαίρι για να έχουμε ε, κατευθυντήριες γραμμές για την εξωτερική δράση και το εξωτερικό μέσον ε, χρηματοδότησης πριν από το τέλος του έτους. Πιστεύουμε λοιπόν ότι μπορούμε να προωθήσουμε έναν ουσιώδη διάλογο σε ένα πρόωρο στάδιο με την Κομισιόν και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν και οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Ως προς τα διδάγματα που αντλήσαμε, ας δούμε την λειτουργία του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας, του DCI, με βάση τον δημοκρατικό έλεγχο και τις ομάδες εργασίας, Έχουμε ένα πλούτο πληροφοριών για τις αδυναμίες και τα θετικά σημεία της εφαρμογής. Το DCI, ο Μηχανισμός Αναπτυξιακής Συνεργασίας, εστιάζει την προσοχή στην εξάλληψη της φτώχειας και των αναπτυξιακών στόχων, έτσι ώστε να δούμε πώς θα αναπτυχθεί η πολιτική μας για την Ασία και τη Λατινική Αμερική. Όλα τα θεματικά προγράμματα ήταν σημαντικά, αν και εκφράσαμε μεγάλες ανησυχίες ως προς τις ε, προτεραιότητες και τη θεματική στρατηγική για θέματα μετανάστευσης. Το 100% της χρηματοδότησης και το 90% των θεματικών προγραμμάτων θα πρέπει να ε, εντάσσονται στους μηχανισμούς αναπτυξιακής συνεργασίας. Η Επιτροπή αναγνώρισε αυτή την ανάγκη προτείνοντας ε, συγκεκριμένους μηχανισμούς για τις αναδυόμενες χώρες με βάση τον ε, κανονισμό ICI+ το 20% δαπανών στην υγεία και την εκπαίδευση μέχρι το 2009 που είχαμε θέσει αποτελεί ένα βασικό σημείο αναφοράς για το Κοινοβούλιο. Χρειαζόμαστε μια εξειδικευμένη έκθεση για να δούμε πώς ε, τηρήσαμε αυτούς τους στόχους με μια κατανομή στον τομέα της εκπαίδευσης και της υγείας. Γιατί χρειάζεται ένα σχολείο, αλλά χρειάζεται και μια οδική αρτηρία που να οδηγεί στο σχολείο Χρειαζόμαστε λοιπόν μία ε, ολιστική προσέγγιση. Διαδικαστικά το εγχείρημα του δημοκρατικού ελέγχου διευκόλυνε έναν επικοδομητικό διάλογο με την Κομισιόν. Το μεγάλο πρόβλημα με το μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας είναι το γράμμα του κανονισμού αλλά η ερμηνεία του. Υπάρχουν, υπάρχει τάση στα κράτη-μέλη να θεωρούν το DCI σαν έναν άλλο μηχανισμό για να προωθήσουμε τις κοινέ αξίες σε άλλες χώρες. Όμως, η αναπτυξιακή συνεργασία και αυτός ο μηχανισμός προωθεί τα συμφέροντα των πιο περιθωριακών πληθυσμών αυτού του πλανήτη. Άρα, επικρίναμε τον προγραμματισμό ο οποίος δεν εστιάζεται στην βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλληψη της φτώχειας, και την διαβούλευση των εμπλεκομένων. Επίσης, τα Εθνικά Κοινοβούλια και η Κοινωνία των Πολιτών δεν συμμετείχαν σε αυτό το διάλογο. Ως προς το μέλλον, ποια είναι τα διδάγματα. Οποιοδήποτε ξεχωριστός μηχανισμός που σχετίζεται με τις αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να εξοπλίζεται από πλευράς ε, χρηματοδότησης, έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα στόχο 0,7% ε, του GNI μέχρι το 2015, δηλαδή μέσα στα πλαίσια του πολιετούς ε, προγράμματος, το οποίο θα πρέπει να αυξηθεί χρηματοδοτικά. Ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να βασιστεί στο άρθρο 208 της Συνθήκης της Λισαβόνας σε σχέση με την εξάλληψη της φτώχειας. Επίσης, η χρηματοδότηση των γεωγραφικών προγραμμάτων θα πρέπει να βασίζονται στον μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας στρίκτο σένσου μέσα στα πλαίσια των DCI, του DCI, δηλαδή του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας. Με βάση αυτό τον μηχανισμό χρειάζεται καλύτερο benchmarking από το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν. Σας μίλησα για την επιστολή του Υφυπουργού, του αναπληρωτή Υπουργού Άντριου Μίτσελ. Δεν θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό. Θα πρέπει να ορίσουμε αυτό αυτή τη στοχοθέτηση με βάση μια περιφερειακή βάση. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένες ε, πληροφορίες για να ξέρουμε κατά πόσο ανταποκρινόμαστε σε αυτή τη στοχοθέτηση. Επίσης να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία έτσι ώστε να μπορούμε να αντιδρούμε στις επερχόμενες ε, αλλαγές και ο μηχανισμός θα πρέπει να καλύπτει όλες τις αναπτυξιακές χώρες έτσι ώστε να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε προγράμματα για αναδιόμενες χώρες και χώρες μέσου εισοδήματος. Ως προς τις διαδικασίες είδαμε ότι ο μηχανισμός αυτός, ο DCI, ο μηχανισμός αναπτυξιακής συνεργασίας έχει μεγαλύτερη επίπτωση στα, ως προς τα προγράμματα στρατηγικής. Μας ενδιαφέρουν τα ενεξελίξη προγράμματα έτσι ώστε να δούμε και θέματα εξωτερικής πολιτικής και εξωτερικής συνεργασίας. Θα πρέπει λοιπόν η ΕΕΔ να προωθήσει αυτά τα προγράμματα και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να προωθήσει τις κατεξουσιοδότηση πράξης μέσα στα πλαίσια της συνθήκης της ε, ε, Λισαβόνας αυτή η συζήτηση συνεχίζεται έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να μπορέσει να προασπίσει αυτή την στοχοθέτηση υπέρ των φτωχών και των φτωχότερων στρωμάτων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπέρμαν έχει το λόγο. Και σύντομα κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για πραγματικά θαυμάσιο έγγραφο. Δεν έχω άλλες ερωτήσεις εκτός από μία αλλά δεν έχει ε, κριτικό χαρακτήρα. Θεωρείτε ότι με τον μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας εκμεταλλεύεται παρκώς η Ευρωπαϊκή Ένωση την συλλογική ισχύ των 27 χωρών μελών, δηλαδή το, την πολιτική βαρύτητα που μπορούμε να προσδώσουμε στο μηχανισμό αυτό που εκπροσωπεί ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να είμαστε δωρητής αντί να είμαστε εκπρόσωπος συλλογικά της προσπάθειας των χωρών μελών, δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να έχουμε μια ισχυρή φωνή στις αναπτυξιακές πολιτικές ως Ευρωπαϊκή Ένωση και να εκμεταλλευτούμε την πολιτική μας ισχύ δίνοντας περισσότερο βάρος σε ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία, ε, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των πιο ευαίσθητων χωρών. Δεν επικρίνω τις θεματικές επιλογές που έχετε κάνει, ούτε θα ζητούσα κατάργησή τους και καλά και βέβαια θα ε, ζητούσουμε να συνεχιστούν οι προσπάθειες αυτές, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να δώσουμε περισσότερη έμφαση στα πλεονεκτήματά μας. Αυτό πιστεύω ότι είναι απαραίτητο. Τι νομίζετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εκπροσωπεί ο κύριος Ντερόσα. Ευχαριστώ και σας κύριε Πρόεδρε και τον κύριο Μίτσελ για την έκθεσή του. Είναι χρήσιμο όντως να εξεταστεί η κατάσταση και να συναχθούν συμπεράσματα. Υπάρχει μια σύγκριση απόψεων συνολικά για τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα. Θεωρώ πάντως ότι θα ήταν σκόπιμο να μπορέσει να χρησιμοποιήσει κανείς την έκθεση με τρόπο πολύ πιο ενεργό. ερχόμενος στα διάφορα κεφάλαια της εκθέσεως, άκουσα βεβαίως τον κύριο Μίτσελ, να λέει ότι η πολιτική αναπτύξεως δεν είναι φτιαγμένη για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η, συνένεση, η Ευρωπαϊκή Συνένεση εν προκειμένου είναι αρκετά σαφής. Με την έννοια ότι η πολιτική ανάπτυξη εξυπηρετεί την προώθηση των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και βέβαια την πρόθεση ενός κόσμου πιο με μεγαλύτερη ισότητα, με λιγότερες συγκρούσεις, λιγότερες ανισότητες, λιγότερη φτώχεια, που και αυτό εξυπηρετεί έμεσα και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ε, μια σταθερότητα, μια ειρηνική ανάπτυξη. ώστε να μην φανεί ότι η πολιτική ανάπτυξη είναι μια ανθρωπιστική πολιτική, που αυτή βέβαια είναι πιο περιορισμένη. Έχει το νόημα να διασώσει ζωές σε μια συγκεκριμένη περίοδο για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ενώ εδώ μιλούμε για μια πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των εξωτερικών της σχέσεων και να είναι ένα, αν όχι το πιο σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής αυτής, απέναντι σε ορισμένες ε, αναπτυσσόμενες χώρες. Σε ό,τι αφορά τα συναγόμενα συμπεράσματα ή διδάγματα, ας εξετάσουμε ποιες, ποια ήταν οι περιορισμοί του ε, μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας ε, με διάθεση 100% των πόρων στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια βλέπουμε συχνά να είμαστε αντιμέτωποι καταστάσεων όπου απαιτείται επίδειξη κάποιας ευελιξίας. Χάρη στο ότι μπορέσαμε να επενδύσουμε τον μηχανισμό ειρήνευσης στην Αφρική για την αντιμετώπιση συγκρούσεων εκεί όπου τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούσαν άμεσα να ε, αναμειχθούν έδειξε, αλλά καθώς επίσης και άλλα παραδείγματα όπως η Food Facility και άλλα, δείχνουν την ανάγκη να υπάρχει ένας μηχανισμός στο μέλλον, να υπάρχει μια προβλεψιμότητα και αυτό είναι σημαντικό και για όλους τους εταίρους μας που βρίσκονται σε κανονική κατάσταση. Από την άλλη μεριά να υπάρχει επαρκής ευκαμψία η ευελιξία ώστε να αντιμετωπίζουμε τις ανάγκες ενός κόσμου που αναπτύσσεται με ταχύτητα και οι πρόσφατες εξελίξεις ε, στο νότιο μέρος της Μεσογείου ε, α, μου κάνετε νόημα ότι θα πρέπει να συντομεύω καλώς ολοκληρώνοντας έχω να πω το εξής ο Επίτροπος έκανε ήδη μια παρέμβαση ενώπιον της ε, Επιτροπής με τις ιδέες αυτές. Είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε με τον κύριο Μίτσελ για να δούμε με, σε ποιο μέτρο μπορούμε να κάνουμε την έκθεση αυτή χρήσιμη και για τη μελλοντική εφαρμογή του μηχανισμού αναπτυξιακής συνεργασίας. Ο κύριος Ντέβα ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου. Ο κύριος Μίτσελ στην επιστολή του λέει ξεκάθαρα το εξή. Τα αποτελέσματα δεν έχουν ε, γίνει μόνο από τον Βρετανικό λαό, αλλά και υπέρ του Βρετανικού λαού. Η δημιουργία δηλαδή ενός ε, πιο ευημερούντος και πιο σταθερού κόσμου, το οποίο θα οδηγήσει σε ασφάλεια και της δικής μας χώρας και από το οργανωμένο έγκλημα και από μεταδοτικές ασθένειες κλπ. Και γι' αυτό η ιστορική απόφαση να αυξηθούν τα επίπεδα σε 0,7% του ΑΕΠ δεν είναι μόνο ηθικά. Ε, θα μας μεταναφέρετε πάλι όλη την Καινή Διαθήκη, λέει ο κ. Δεν κάνουμε εδώ ανάπτυξη επειδή είμαστε υποχρωμένοι ηθικά. Το κάνουμε και για να διατηρήσουμε ασφαλέστερη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Μίτσελ ας ολοκληρώσει. Νομίζω ότι η, παρα, παραπομπή του κύριου Ντέβα ήταν για τον άλλο κύριο Μίτσελ που ανέφερα προηγουμένως, όχι για μένα, τον Υπουργό δηλαδή. Τώρα, κοιτάξτε κύριε Πρόεδρε, για τα όσα είπε ο Επίτροπος. Αν πάρουμε το ευρύτερο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαϊκών χωρών μελών και πούμε ότι είμαστε οι μεγαλύτεροι δωρητές, ορισμένες χώρες ε, ε, ε, επιδιώκουν πρόθεση των δικών τους στόχων και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα εδώ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Έρχομαι σε αυτά που είπε ο κύριος Μπέρμαν προηγουμένως. Υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερη συνοχής στον τρόπο που διεξάγουμε τις υποθέσεις μας, αλλά με μεγαλύτερη συνοχή θα μπορούσαμε να διαθέτουμε και 6 δις παραπάνω τον χρόνο, είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό βέβαια το επιχείρημα μπορεί να συνεχίζεται επάπειρον. Ίσως πρέπει τώρα, στα μισά της θητείας της παρούσας Βουλής, να ζητήσουμε μια κοινή συνεδρίαση με το Συμβούλιο Υπουργών Ανάπτυξης σε ισομερή βάση. 27 βουλευτέ και 27 υπουργοί. Να δούμε από πού μπορούν να βρεθούν τα 6 δισεκατομμύρια. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό κάθε εβδομάδα. Αλλά αφού πρόκειται για διαδικασία συνδιαλλαγή, α το κάνουμε αυτό. Είχα συναντηθεί με το Συμβούλιο όταν ήμουν και εισηγητή για την Emergency Food Facility. Α συναντηθούμε μαζί του να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη συνοχή. Αυτό νομίζω ότι θα ήταν και χρήσιμο και σωστό, όπως άλλωστε είπε ο Τάις Μπέρμαν. Η πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε στο 13 της ε, ημερήσιας διάταξης. Πρόταση συστάσεως του Συμβουλίου για την 60 έκτη ε, σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών. Η κυρία Στρίφλερ είναι ε, η εισηγήτριά μας. Έχει αμέσως τον λόγο. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, Καλούμαστε να συμβάλλουμε με την ομοδότησή μας ε, στην έκθεση ΑΦΕΤ για τις συστάσεις για την 66η έκθεση Σύνοδο, όπως Έχουμε τα εξή θέματα. Στόχου χιλιετία για την ανάπτυξη, λιγότερο αναπτυγμένε χώρε, αποτελεσματικότητα τη βοήθεια και δικαίωμα στην ανάπτυξη. Και θα πρότεινα στη συνέχεια να προσθέσουμε και θέματα που έχουν να κάνουν με την ανθρωπιστική βοήθεια που θα απασχολήσουν την προσεχή διάσκεψη των ΗΠΑ. Η στόχη της χιλιετίας συγκεκριμένα ε, νομίζω ότι μπορούν να υλοποιηθούν με βάση τους τέσσερις εξής ανανέωση των δεσμεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο και της κοινή δέσμευση για σεβασμό των στόχων της χιλιετίας για το 2015 δεύτερον να πρέπει να ξανασυζητήσουμε πώς μετά το 2015 η δέσμευση διεθνούς κοινότητας για τη βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να ε, πραγματοποιηθεί και πώς μπορούν να αποτελέσουν αυτοί οι στόχοι βάση για την πλήρη εξάλληψη της φτώχειας στον κόσμο. Τρίτον, να στηρίξουμε την χρηστή διακυβέρνηση και να λάβουμε μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής, να ε, βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών πάλι με προοπτική του στόχου χιλιετίε. Όπω ξέρετε, λιγότερο αναπτυγμένε χώρε ε, θα συζητηθούν με τέταρτη διάσκεψη στην Κωνσταντινούπολη, όπω υπόθηκε και νωρίτερα. Και η Επιτροπή Ανάπτυξη θα έχει ιδιαίτερα ε, την εκπροσώπησή τη εκεί. Στόχο έχουμε λοιπόν να δώσουμε προτεραιότητα στα εξή ζητήματα που πρέπει να προβληθούν, επιστηστική ασφάλεια, γεωργία υποδομές, ε, capacity building, οικονομική ανάπτυξη με συμμετοχή των πάντων, νέες τεχνολογίες και κοινωνική και ανάπτυξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Θα πρέπει επίσης να υποστηριχθεί, να εξασφαλιστεί μάλλον δυνατότητα για την λειτουργία των μηχανισμών ελέγχου και διαρκού παρακολούθησης με προοπτική την εφαρμογή του προγράμματος των μόνων Αθηνών για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες ενώπιση της νέας δεκαετίας. Και επίσης στη διάσκεψη θα πρέπει να συζητήσουμε τη μετατροπή του προγράμματος για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας ώστε να μετατραπεί αυτό σε πρόγραμμα για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης με βάση το πρόγραμμα της Άκρα και με πλήρη δέσμευση των κοινοβουλίων της κοινωνίας των πολιτών και των ε, τοπικών αρχών. Το δικαίωμα στην ανάπτυξη είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που θα πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντο σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι το δικαίωμα στην ανάπτυξη. Εφέτο, όπω σα είπα, χαιρετίζουμε την 25η επέτειο τη διακήρυξη των ΗΠΑ για το δικαίωμα στην ανάπτυξη και προκειμένου να ε, εξασφαλιστεί η διατήρηση και ο σεβασμός αυτής της διακήρυξης έχουμε θεσπίσει ε, μια task force για τη θέσπιση του δικαιώματο του 2004 μαζί με το σχετικό συμβούλιο. Παράγραφό 1, εδάφιο 1 τη εκήρυξη πρόκειται η, η ανάπτυξη είναι παλωτρίο το δικαίωμα κάθε ανθρώπινου όντως, κάθε έχει δικαίωμα να συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ανάπτυξη προκειμένου να υλοποιούνται όλες οι προσδοκίες των ανθρώπων και να αποφυλείται ο καθένα από την ανάπτυξη. Και άρα η Task Force υψηστού επίπεδου του 2004 πιστεύω ότι θα πρέπει να βοηθήσει στην ουσιαστική υλοποίηση της, ε, του δικαιώματο στην ανάπτυξη και θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αναγνωριστεί η σημασία του δικαιώματο αυτού, η εγγραφή του στην Οικουμενική Διακήρυξη και του μηχανισμού προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών υπό την αιγύδα των ΗΠΑ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Κόρτε Λάστρα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Στίφλερ, για την εξαιρετική αυτή έκθεση. Εγώ συμμερίζομαι πολλά από τα σημεία που προαναφέρθηκαν. Καταρχήν θα πρέπει να ανανεώσουμε τη δέσμευση αυτή σε σχέση με τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας και τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Να αυξήσουμε την αναπτυξιακή βοήθεια λοιπόν. Συμμεριζόμαστε αυτούς τους τέσσερις, τέσσερις στόχους και τη χρηστή διακυβέρνηση καθώς και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την φοροδιαφυγή και να υποστηρίξουμε την πρόληψη διαφορών. Ως προς καινοτόμους μηχανισμούς νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι χρηματοοικονομικές δράσεις σε πρώτη φάση που θα ορίσουμε και να θέσουμε ε, ορισμένες προτεραιότητες για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε με τα Ηνωμένα Έθνη και δεν πρέπει να ξεχνάμε και για τις χώρες μέσω εισοδήματος, διότι δεν θα πρέπει να τις αγνοήσουμε μέσα στα πλαίσια της καταπολέμησης της φτώχειας. Επίσης, θα πρέπει να προσδώσουμε σημασία στη μείωση διαφορών και ανισοτήτων για να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια. Να δώσουμε μεγάλη, μεγαλύτερη σημασία στην κατάσταση των γυναικών, διότι πλήττονται περισσότερο από την ε, φτώχεια. Θα πρέπει να προωθήσουμε λοιπόν την ισότητα ευκαιριών και να είναι πιο συνεκτικές οι πολιτικές μας, οι αναπτυξιακές μας πολιτικές και πιο συνεπείς. Το λόγο έχει η Επιτροπή, ο κύριος Πίτερ Κρέγκ Μακουέιντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ως προς την προετοιμασία της θέσης μας για την 66η διάσκεψη, έχουν γίνει, οι, οι, πρώτες συζητήσεις θα γίνουν στις 15 Μαρτίου στα Ηνωμένα Έθνη. Θα πρέπει να προσδώσουμε μεγάλη σημασία στους αναπτυξιακούς στόχους και στις ΛΑΧ. όπως αναφέρεται και στην έκθεση Στρίφλερ. Επίσης, έχουμε μία, θα πρέπει να έχουμε μία σωστή προσέγγιση η οποία να μην είναι θεωρητική υφής. Βεβαίως θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία και στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως ορίσαμε στην Σύνοδο για τις ΛΑΧ πέρσι μέσα στα πλαίσια των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Επίσης θα πρέπει να έχουμε έχουμε καλύτερους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. Ο κύριος Κορ, όπως είπε και ο κύριος Κόρτες Λάστρα, θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στις ΛΑΧ και τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας μέσα στα πλαίσια της χρηστής διακυβέρνησης, της καταπολέμησης της διαφθοράς και της σημασίας των γυναικών και μιας συνεκτικής και συνεπούς πολιτικής μέσα στα πλαίσια της συνέλευσης, της Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών μετά από τα συμπεράσματα της Κωνσταντινούπολης. Η κυρία Στίφλερ έχει το λόγο για να συνοψίσει. Θα λάβω υπόψη τις προτάσεις του κυρίου Κόρτες ως προς τον ε, μηχανισμό, τον καινοτόμο μηχανισμό χρηματοδότησης, να επιμείνουμε περισσότερο στις γυναίκες και δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Συμφωνούμε ως προς το περιεχόμενο. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ως προς το περιεχόμενο. Η κυρία Στίφλερ αναλαμβάνει την Προεδρία για το τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Euh, euh, Παίρνουμε στο σημείο 14 της μέρη σας διάταξης το νέο πρωτόκολλο μέσα στα πλαίσια της αλίας και της χρηματοοικονομικής αντιστάθμισης όπως ε, ε, αναφέρεται στην Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δημοκρατίας των Σεϊχελών. Δίνω το λόγο στον εαυτό μου. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίο το βρίσκω αυτό. Θα είμαι πολύ σύντομη. Τα συμβαλόμενα μέρη θα πρέπει να προωθήσουν μία υπεύθυνη αλία με βάση την αρχή της μη διάκρισης μεταξύ των διαφόρων αλλιευτικών στόχων στα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας των Σεϊχελών. Το χρηματικό αντιστάθμιμα αφορά 16.800.000 ευρώ μέσα στα πλαίσια των συνολικών αλλιευμάτων και αν, αν είμαστε πάνω τις 52.000 τόνους, τότε θα πρέπει να υπάρχει ένα επιπρόσθετο ποσό ανατόνο εκ των 65 ευρώ. Όταν υπερβαίνουμε τα αντίστοιχα ποσά στο διπλάσιο, δηλαδή όταν η υπέρβαση είναι πάνω του διπλασίου, τότε αυτό έχει αντιστάθμισμα το επόμενο έτος. Ο επιμερισμός αυτών των πόρων αφορά αποκλειστική αρμοδιότητα των Σεϊχελών. Άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιοι ευεργετούνται από αυτούς τους πόρους. Άρα η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης θα πρέπει να είναι ένα ε, νόμιμο και θεμητό μέσο, αλλά θα πρέπει να επιτρέπει την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των θαλασσίων χώρων. Το χρηματοοικονομικό αντιστάθμο που θα αφορά τον Ευρωπαίο φορολογούμενο θα πρέπει να προωθείται προς τους αναπτυξιακούς στόχους υπέρ των ε, αλληλευτικών κοινοτήτων μέσα στα πλαίσια της κατάρτισης, της ασφάλειας στη θάλασσα και τη δημιουργία νέων θέσεων ε, εγχώρια εργασίας. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ε, θέση σε ισχύ της συμφωνίας. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια για τα συνολικά αλλιεύματα. Ο μηχανισμός θα πρέπει να βελτιωθεί και θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι καταπολεμούμε την διαφθόρα και η κυβέρνηση θα πρέπει να βελτιώσει την ε, ποιότητα ζωής των εγχώριων αλλιέων. Επίσης, θα πρέπει να τηρήσουμε τις περιφερειακές προδιαγραφές και να έχουμε σύνταξη ενδιάμεσων εκθέσεων που θα διαβάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Κέλλερ ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ σύντομα. Πρέπει πιστεύω να υπάρχει ένα νότο επίπεδο για την ε, περιφέρεια ολόκληρο, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα αποδομητικό είδο, τον τόνο δηλαδή, ο οποίο αποδημεί και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να υπάρχει ανώτατο επίπεδο μόνο για τις Αιχέλες, αλλά επιπλέον ε, προσθήκη ποσού, επιπλέον καταβολή ποσού για ολόκληρη την περιφέρεια και όχι μόνο για τη χώρα. Σε περίπτωση Υπερβολικό λεύματο. Και ερώτηση προ την Επιτροπή, τι κάνει η Επιτροπή για να περιορίσει επιπτώσεις τη όλο και, ενισχυόμενη όλο των λεγόμενων fishing aggregating devices που σημαίνουν ουσιαστικά περισσότερη αποτελεσματικότητα στην αλία, δηλαδή συλλαμβάνονται περισσότερα ψάρια. Τι κάνετε για να καταπολεμήσετε αυτό το φαινόμενο. Alors, je vais passer la parole à la Commission à Monsieur. Δίνω το λόγο στον κύριο Αλεξάνδρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύντομα παρακαλώ, διότι σε πέντε λεπτά θα χάσουμε τους ερμηνείς. Έχετε τρία λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και κυρία Συγγήτρια. Θα ήταν θαύμα να μπορούσα να σας τα ε, λύσω όλα τα προβλήματα μέσα σε τρία λεπτά. Άκουσα μεγάλη ε, μεγάλο θαυμασμό την ε, έκθεσή σας, την παρουσίαση αυτή συνοπτική. Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση, σε ορισμένα σημεία μπορώ να συμφωνήσω. Και για να είμαι ε, αντικειμενικός θα πρέπει επί τη ευκαιρία να επανέλθω σε ορισμένα σημεία, για όσο πιο πολλές πληροφορίες. Και για να δώσω την απάντηση στην κυρία Κέλλερ, συμφωνούμε ότι πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια προκειμένου να μην μετέρχονται ορισμένοι αυτές τις ε, μεθόδους αλίας των FAD, Fisheries Aggregating Devices, που ορισμένοι μπορεί να θεωρούν καταστροφικές. Σε περιφερειακό επίπεδο λοιπόν και από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σε θέματα των νοηδών του Ινδικού ωκεανού εργαζόμαστε και κάθε απόφαση σε περιφερειακό επίπεδο έχει και την, ε, το αντίστοιχό της, αντικατοπτρίζεται δηλαδή στις συμφωνίες με τα τρίτα κράτη. Αυτή είναι η απάντηση για την περιφερειακή πτυχή. Για τον προσδιορισμό ενός του ορίου, και πάλι σε περιφερειακό επίπεδο, θα επενθυμίσω ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με περιφερειακή συμφωνία. Πρόκειται για διμερή συμφωνία, η οποία λαμβάνει όμως υπόψη την περιφερειακή διάσταση που αναπτύσσει και ουσιαστικά προστατεύει πάλι η Επιτροπή των Τονοειδών του Ινδικού Ωκεανού. Ε, και σε τούτου συμφέρον όλων μας και δικό σας και δικό μας και των ΣΥΧΕΛΟΝ για την προστασία αυτών των αποθεμάτων τόνου είναι να υπάρχει μια προσπάθεια συντονισμένη σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά συντονισμένα και με το διμερές, με τη διμερή συμφωνία. Υπενθυμίζω ότι η Σεϊχέλες είναι ένα εκ των συμβαλωμένων μερών, αλλά από τα πιο δυναμικά και δραστήρια, με τη θετική έννοια του όρου, μέρη της ε, προσπάθειας για την προστασία των αλληλευτικών πόρων ε, στο χώρο που καλύπτει η σύμβαση OI, η Περιφερειακή δηλαδή Επιτροπή Διαχείρισης των Πόρων. Και αν περισσεύουν δύο λεπτά, εσεί θα μου πείτε πρόεδρε, θα ήθελα να δώσω κάποιες διευκρινήσει σε ορισμένα σημεία της ε, ομιλία σας που θεωρώ σημαντικά και πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσω απαντήσει, αλλά θα μου πείτε εσεί. ενάμιση λεπτό. Καλώ θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. πρόεδρε. Το νέο αυτό πρωτόκολλο το διαπραγματευτήκαμε το 2010. Και πριν από την ε, εκκίνηση μεταρρύθμιση την εξωτερική διάσταση, ασχοληθήκαμε ήδη το 2010 με την αναγκαιότητα ε, να προσαρμοστούν ορισμένε έννοιε κλειδί του πρωτοκόλου, φέρει πίν και υπογραμμίζει ιδιαίτερο στο γεγονό ότι στο οικονομικό αντιστάθμισμα ξεχωρίσαμε δύο ε, κατηγορίες. Ένα είναι η πρόσβαση και είπαμε ότι η πρόσβαση, το τμήμα που έχει να κάνει με την πρόσβαση προσδιορίζεται με βάση τη βούληση του τρίτου κράτους, όμως το διμερές τμήμα εξαρτάται από τον προγραμματισμό και τη δουλειά που θα πρέπει να επιτελέσουν στην Μικτή Επιτροπή οι δύο πλευρές με παρακολούθηση τακτική ώστε να εξασφαλίσετε τη τήρηση των στόχων και η επιτευξή τους και εδώ ακριβώς κυρία Πρόεδρε συμφωνούμε ιδιαίτερος προκειμένου να εξασφαλιστεί ουσιαστικός αντίκτυπος επίπεδο στήριξης της ε, βιοτεχνικής αλίας που είναι πολύ σημαντική για την ε, ε, διατροφή σε πρωτεΐνες του πληθυσμού. Και εδώ περνούμε τώρα στην ρήτρα άρσης του πρωτοκόλου σε περίπτωση παραβίας ανθρωπινών δικαιωμάτων. Καιροτομία που εισήχθη το 2010, όλα τα πρωτόκολλα που διαπραγματευόμαστε από το 2010 και εξής προβλέπουν μια ρήτρα άρσης και όπως είπα πρόκειται για πρώτη φορά που το έχουμε αυτό, εάν διαπιστωθούν προβλήματα στα ανθρώπινα δικαιώματα, έρεται η λειτουργία της συμφωνίας, η ισχύ συμφωνίας και του πρωτοκόλου Και για τα ε, κονδύλια που έχουν να κάνουν με τη διμερή συμφωνία, εάν από τον ένα χρόνο στον άλλο δεν τηρούνται ε, τα συμφωνημένα ποσά ή ποσότητε καλύτερα, η Επιτροπή μπορεί να άρει τη λειτουργία του διμερούς κομμάτιου της συμφωνίας. Και αυτό είναι το καλύτερο, ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε αποτελεσματικά με το τρίτο κράτος, ώστε οι, κοινοί, οι κοινώς στόχοι να επιτευχθούν. Πρόεδρε, πιστεύω να ήμουν αρκετά σύντομο και να συνέβαλα στις συζητήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινήσεις αυτές. Δεν θα ξαναλάβω το λόγο, γιατί πρέπει να βιαστούμε. Επιτρέψτε μόνο να υπενθυμίσω ότι έχουμε προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών στις 12 το μεσημέρι 4 Μαρτίου και ψηφοφορία στις 22 Μαρτίου. Και ένα τελευταίο σημείο, το δημοκρατικό έλεγχο του προγραμματισμού στο πλαίσιο της νομοθεσίας που διέπει την αναπτυξιακή πολιτική, με τον κύριο Γκέρενς, πρόεδρο της ομάδας εργασίας Περιθμών ΔΕΛΤΑ, ο οποίος είχε την καλοσύνη να αντικαταστήσει τον κύριο Τσιρολιά. Το λόγο έχει ο κύριος Γκέρενς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να αντικατοπτρίσω τη θέση του κυρίου ε, Τιρολιέν. Ε, συμφωνεί εμπολής με την Κομισιόν Ζητούμε λοιπόν από την Επιτροπή Άτιο Ρεωνέο για σας να μην ε, αρνηθείτε τη στρατηγική του 2011-2013 ως προς το, τα προγράμματα τα οποία δεν έχουν κρατικό χαρακτήρα. Γι' αυτό θα θέλαμε να λάβετε υπόψη αυτά τα προγράμματα μέσα στα πλαίσια των ε, θεματικών ενωτήτων. Ως προς τις έξι συστάσεις, μετά από την ανάγνωση του προγράμματος στρατηγικής, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο μόνο σημείο. Πρόκειται για το γεγονός ότι μετά από τρία χρόνια πολλοί θεώρησαν, από τρία χρόνια λειτουργίας θεώρησαν θα, πολύ ενδιαφερόμενοι ότι θα πρέπει να υπάρχει πιο στενή συνεργασία μεταξύ των μη κρατικών τοπικών φορέων και των τοπικών αρχών. Διότι οι ανάγκες των τοπικών αρχών είναι πολύ διαφορετικές από έναν μη κυβερνητικό οργανισμό. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν ορισμένες διευθετήσεις για να λάβουμε υπόψη αυτές τις ιδιαιτερότητες. Όμω, όπως είδαμε στον ε, διαρθρωμένο διάλογο, η μέθοδος διαχείρισης θα μπορούσε να οδηγήσει σε τριβές μεταξύ μη κυβερνητικών και τοπικών αρχών. Για να μην υπάρχει λοιπόν αυτός ο άλογος ανταγωνισμός, θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να σκεφτεί σοβαρά το όλο ζήτημα, όπως κάνει πάντα, μέσα στα πλαίσια του ΙΣΕΝΤΕ 2014 έτσι ώστε να προωθηθούν διαφοροποιημένες προτάσεις. Και τρίτο σχόλιο και τελευταίο, η δική μας Επιτροπή ζητά την διαβούλευση με τους επιτόπιους φορείς όπως αναφέρουν τα άρθρα 19 έως 33 της Σύμβασης του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, έτσι ώστε να επέλθει μια βελτίωση. Εγώ συμμετέχω πολύ συχνά σε αυτές τις διαδικασίες αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μία μακρογεωγραφική ε, προσέγγιση, όμως οι επιλέξιμες χώρες δεν έχουν δείξει ενδιαφέρον μέχρι τούδε, γι' αυτό θα πρέπει να επιδείξουμε μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την συμμετοχή των επιτόπιων φορέων. Γνωρίζουμε τους περιορισμούς, ιδιαίτερα ως προς το ανθρώπινο δυναμικό, που δεν επιτρέπει σε ορισμένε αντιπροσωπείες να επιτελέσουν αυτή την εργασία. Όμως έχει μεγάλη σημασία, διότι μέσα στα πλαίσια κάθε αντιπροσωπείας θα πρέπει να υπάρχει ένας υπεύθυνος για τη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και η Επιτροπή να μας ενημερώνει για την πρόοδο των ε, διαπραγματεύσεων. Αυτά έχει να μας πει ο φίλος Τυρολιέ ο οποίος δεν μπόρεσε να παραστεί σήμερα. Νομίζω ότι για μία φορά ήταν ιδιαίτερα ευγενής με την Επιτροπή. Και ευχαρι... σας ευχαριστώ όλους όσους παρίσταστε, γιατί με παρακολουθήσατε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε κύριε Γκέρενς. Η κυρία Βίλμαν Δεν τολμώ καν να σας πω πόσο χρόνο έχετε στη διάθεσή σας. Θα λάβουμε αυτά τα σχόλια γραπτός, θα τα ξανασυζητήσουμε εν ευθέτω χρόνο. Συμφωνούμε με τα σχόλια, προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη διαδικασία και αυτά τα ολίγα. Θα τα ξαναπούμε για να το συζητήσουμε. Ε, εντάξει, ως προς τα συμπεράσματα. Ε, θα πω στον κύριο Τυρολιέν για την αντίδραση της Κομισιόν, η οποία είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη. Ωραία, κλείνει η διαδικασία δημοκρατικού ελέγχου σε σχέση με τα θεματικά προγράμματα. Μιλάμε για μη κρατικούς φορείς και τοπικές αρχές, την αναπτυξιακή διαδικασία Έχουμε κι άλλο ένα θέμα. Κύρια Κέλλερ, για τη διαδικασία δημοκρατικού ελέγχου, θεματικά προγράμματα, μετανάστευση και άσυλο. Σας ευχαριστώ τους διερμήνες εκ των προτελών Κέλλερ. Για το θεματικό πρόγραμμα μετανάστευσης, ακούσαμε τον κύριο Μίτσελ πριν και την κριτική που άσκησε τα ίδια πράγματα μπορούν να λεχθούν και εδώ. Έχουμε κάνει ανταλλαγή απόψεων με διάφορους εκπροσώπους της Επιτροπής, έχουμε λάβει και έχουμε αποστείλει ερωτήσεις και απαντήσεις. Το συμπέρασμα εν τέλει είναι, όπως είπε ο κύριος Μίτσελ, και το πρόγραμμα αυτό εστιάζεται πολύ στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι τόσο τις αξίες, αλλά τα συμφέροντα. Κυρίως ό,τι αφορά την διαχείριση μεταναστευτικών ροών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι μεταναστευτικών ροών από νότο σε νότο. Είναι δύσκολο να αποδειχθούν ορισμένα από τα στοιχεία αυτά. Η σχέση επίσης με την φτώχεια όταν μιλούμε και για εκπαίδευση ε, μεθοριακών φρουρών για τον εντοπισμό πλαστογραφημένων διαβατηρίων και ούτω καθεξής. Αυτά επίσης είναι λίγο δύσκολα. Τα ίδια προβλήματα λοιπόν που είπε ο κύριος Μίτσελ και πριν. Έχουμε επίσης εδώ το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός προκειμένου είναι ασαφής. Για τι θεματικές προτεραιότητες το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι για κάθε θεματική προτεραιότητα θα είναι μεταξύ 10 και 20% των κονδυλίων που έχουν ε, δεσμευτεί για αυτές. Είναι πολύ ασαφής αυτή η ένδειξη. Εδώ λοιπόν διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Υποτίθεται ότι θα έχουμε ένα προϋπολογισμό λεπτομεριακό, δεν ξέρω τι μπορείτε να πείτε εδώ. Έχουμε και την κατάσταση ότι τα κονδύλια, δηλαδή ο ίδιος ο συνολικός προϋπολογισμός για τα θέματα αυτά είναι πολύ περιορισμένος, ενώ τα έργα είναι πολύ ευραία. Υπάρχουν και πολλές προτεραιότητες και πολλά θέματα που πρέπει να συζητηθούν πώς είναι δυνατόν να γίνουν όλα αυτά με τόσο λίγα χρήματα διαθέσιμα. Εν τέλει, λάβαμε απαντήσεις όπως είπα ότι η ένδειξη θα είναι μεταξύ 10 και 30%. Είπα ότι είναι πολύ ασαφές αυτό. Είναι πολύ δύσκολο αν όχι αδύνατον να καθοριστεί οτιδήποτε πιο συγκεκριμένο. Στο τέλος ε, λοιπόν της γραφής ως εισηγήτρια προτείνω να μην ε, προβληθεί ένσταση στο θεματικό πρόγραμμα για την ώρα, αλλά να θέσουμε τα θέματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στην έκθεση του κ. Μίτσελ, αλλά και, και για μένα το ίδιο ισχύει. Να τα λάβουμε λοιπόν υπόψη αυτά, διότι είναι σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όχι μόνο σε αυτό το θεματικό πρόγραμμα αλλά και σε άλλα και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε αλλιώς δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε τον δημοκρατικό μας ρόλο ελέγχου δηλαδή της εφαρμογής των στρατηγικών προγραμμάτων. Monsieur Pennington, si vous voulez, quelques διεξαγάγαμε ενδιαφέρουσα συζήτηση και χαιρόμαστε για τα σχόλια της κυρίας Κέλλερ. Ελπίζω ότι οι περαιτέρω πληροφορίες που διαθέσαμε θα δείξουν ότι λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις ανησυχίε του Κοινοβουλίου. Αυτό ήταν ενδιαφέρον για μας να δούμε πώς δηλαδή ερμηνεύεται τις πέντε προτεραιότητες των θεματικών αυτών προγραμμάτων και κυρίως όταν τα περισσότερα κονδύλια γίνονται μεταξύ ε, ε, γίνονται με ε, προσκλήσεις εκδηλώσεων ενδιαφέροντος. Στοχεύουμε ωστόσο να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε κάθε μια από τις προτεραιότητες αυτές και όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα ελπίζω θα μπορέσουμε να σας το αποδείξουμε. Ευχαριστώ. Κυρία Κέλλερ, θέλετε να ξαναμιλήσετε. Ναι, πρόκειται στα τέλη Μαρτίου να συντάξουμε ψήφισμα όπου θα περιλαμβάνουμε τις δυσκολίες και τα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει. Η Προεδρεύουσα, σας ευχαριστώ. Ας, θα ε, τότε τα συμπεράσματα την στην επόμενη συνεδρίασή μας. Υπάρχουν διάφορα. Η, συνεδρίαση, η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις Βρυξέλλες στις 22 Μαρτίου από τις 3 έως τις 6.30. Ε, Ολοκληρώνεται το εργασία μας. Σας ευχαριστώ όλες και όλους, καθώς και τις διερμηνείς.